Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Αλλάξαμε βέβαια ε, τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αρχίζουμε με τα σημεία 9 και 10. Ο, στο 9 εισηγητής είναι ο κύριος Τοζανόφσκι. Θα ήθελε να μας κάνει μια εισαγωγή και μετά θα το συζητήσουμε. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο, που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσω, να σας πω μερικά πράγματα για τις εξελίξεις στο, σχετικά με τον Καλλιλέο, μάλλον με το ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης. Θα ευχαριστήσω πρώτα πρώτα την γραμματεία η οποία ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική, μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό εικόνα έχει κανεί σωστή γραμματιακή υποστήριξη όταν πρόκειται για ένα τόσο περίπλοκο θέμα όπως αυτό που συζητείτε ε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, το σχέδιο έκθεσης έχει σαν στόχο να δώσει πληροφορίες <clears throat> και για τον έλεγχο ότι τα δικαιώματα ελέγχου που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ζήτημα αυτό. Επίσης υπάρχουν τροπολογίες η τροπολογία 7 και η τροπολογία 8 είναι σημαντικές ε, νομίζω εδώ για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, μετά ερχόμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο το ανατίθεται στο όργανο αυτό ε, κάποιες εξουσίες ε, λόγω και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν ενδιαφέρει ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να μπορεί να συμμετάσχει και να μπορεί να λαμβάνει μέρος στη διαχείριση. Υπάρχουν εδώ πολύ συγκεκριμένοι κανόνες και ποσοστά που πρέπει να τηρούνται για την απόφαση ε, που παίρνετε κάθε φορά και μετά από πάρα πολλές συζητήσεις δόθηκε ένα 30% στον εκπρόσωπο των, των ψήφων αν θέλετε στον εκπρόσωπο της Κομισιόν ούτως ώστε να μπορεί να παίρνει αποφάσεις κομισιών για σοβαρά θέματα αλλά να μπορούν να μπορούν και τα κράτη-μέλη να αντιδράσουν διότι βεβαίως θέλουμε και τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν ενεργά και να μπορούν να ελέγξουν εντό εισαγωγικών την Κομισιόν, αν θέλετε. Θεωρούμε ότι με το 30% αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Και ελπίζουμε η διαδικασία αυτή να γίνει αποδεκτή. Τρίτο σημαντικό θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η διαπίστευση ή της ασφάλειας αν θέλετε ε, του όλου συστήματος. Η αποτελεσματικότητα ε, ενισχύεται, βελτιώνεται με τις ε, σχετικές προτάσεις και αποφεύγονται παρεξηγήσει, διαδικασίες πολύπλοκες τύπου ε, τροπολογίας κλπ. Ελπίζουμε η διαδικασία που προτείνεται και εδώ για τη διαπίστευση της ασφάλειας να ε, γίνει αποδεκτή. Υπάρχει παρόλα αυτά η τροπολογία επαριθμών 10 ε, σχετικά και αναφέρεται, ζητείται να, με την τροπολογία αυτή να γίνει σαφές ότι είναι ανεξάρτητα και αντικειμενικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος τα μέλη του Συμβουλίου Διαπίστευσης Ασφαλείας. Υπάρχει παρακάτω η τροπολογία 11 για την ε, έγκριση με πλειοψηφία τριών τετάρτων των αντιπροσώπων των κρατών μελών και οι κανόνες αν θέλετε ψηφοφορίας για να μην θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται η συνήθις ειδική πλειοψηφία. Επίσης, Ε, ε, ε, αναφέρεται εδώ στο σχετικό θέμα για την διαπίστευση της ασφάλειας ότι η Κομισιόν πρέπει να παίρνει συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορεί να εγκρίνει κάποια ε, απόφαση διαπίστευσης όμως έχει υποβληθεί σχετικά η τροπολογία 12 ούτως ώστε εάν και εφόσον η απόφαση της Επιτροπής ε, δεν γίνεται αποδεκτή από όλους ε, και δεν λαμβάνεται υπόψη ε, υπάρχει δυνατότητα, δυνατότητα δράσης. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, ιδιαίτερα την ε, Σουηδική Προεδρία η οποία μας βοήθησε και ε, πιστεύουμε ότι ε, βεβαίως η επόμενη συζήτηση θα λάβει μέρο χώρα υπό Ισπανική Προεδρία με την ε, συζήτηση με την Κομισιόν βεβαίως ε, και ελπίζω η Ισπανική Προεδρία να ακολουθήσει τη, το παράδειγμα της Σουηδικής Προεδρίας και ελπίζουμε επίσης ότι θα υπάρχει η από όλου καλή πρόθεση και ενδεχομένως να περάσει το θέμα αυτό μετά την πρώτη ανάγνωση. Είναι πιθανό αυτό τον Ιανουάριο θα έρθω σε επαφή και με τον Σκεώδη εισηγητή ούτως ώστε να συζητήσουμε τις τροπολογίες και να ψάξουμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις τόσο ώστε να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ήδη από τώρα αυτούς που έχουν υποβάλει προτάσεις ή που θα υποβάλουν προτάσεις στο μέλλον για να μπορέσουμε τελικά να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση για αυτό το περίπλοκο τελικά θέμα τη διαχείριση του Γαλιλαίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ρεμέκ, ο σκιώδης εισηγητής, παρακαλώ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις εργασίες του και ε, για τη συνεργασία μαζί μου ως και όδους Θα ήθελα να πω ότι μπορώ να υποστηρίξω το σχέδιο έκθεσης στο σύνολό του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο εισηγητής ε, τόνισε την ε, ανάγκη συνεργασίας με όλους και ε, δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 3 και 8. Εγώ νομίζω ότι θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ του 30% για την Κομισιόν ε, που ήταν 50% και όσον αφορά τώρα την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβουλίο είμαι υπέρ της αντιπροσώπευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκεί ακόμη και αν αυτό δημιουργήσει προβλήματα εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο ουσιαστικά σώσαμε το πρόγραμμα Γαλιλαίο νομίζω λοιπόν ότι δικαιούμεθα να είμαστε παρόντες στο Διοικητικό Συμβούλιο Τώρα από εκεί και πέρα ποιο θα εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θα είναι ευρωβουλευτέ ή όχι, δεν το ξέρω, μπορεί να συζητηθεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Θα ήθελα να πω ήδη εξ ότι ευχαριστώ για τη συνεργασία, γιατί η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή το, το σχέδιο έκθεσης είναι καλό και το 30% που αναφέρθηκε ήδη του συνόλου των ψήφων ε, είναι ε, καλό, συμφωνώ. Όμως για την ε, με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ενημέρωση θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα από αυτά που λέγονται μέχρι τώρα. Ε, Βεβαίω μπορεί να έχει κανεί αμφιβολίες του για το κατά πόσον η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ε, η παρουσία του Κοινοβουλίου ε, οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδιαίτερα σε περίπλοκα θέματα όπως τον Καλλιλέο. Παραδείγματο χάρη ε, για την ε, προκήρυξη διαγωνισμών για το κομμάτι το δορυφορικό υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια αλλά εδώ υπάρχει ακριβώς το πρόβλημα του κατά πόσον θα γίνει ε, χωριστός διαγωνισμός 250 ε, εκατομμύρια ευρώ είναι αυτό για το οποίο συζητούμε ή όχι καταλαβαίνετε τέτοιου είδου προβλήματα δεν ξέρω εάν και εφόσον ε, μπορούν να, γίνουν αντιληπτά από τους εκπροσώπους ε, μας ή όχι και αν αυτό βοηθά στη μεγάλη, μεγαλύτερη διαφάνεια τέλος πάντων δεν είμαι αντίθετος συμφωνώ ότι μπορεί να περάσει και όλα στο θέμα μετά την πρώτη ανάγνωση. Συμφωνώ με όλα αυτά που ελέγχθησαν. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κυρία Νίμπλε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή ε, και εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία μας ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα τον ευχαριστώ λοιπόν για τις ανοιχτές επικοινωνίες που οδήγησαν σε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και στο, στην έκθεση αυτή την οποία υποστηρίζω ε, απόλυτα και φαντάζομαι και η πολιτική μου ομάδα θα την υποστηρίξει. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω όμως. Ζητώ συγγνώμη που θα με ακρηγορήσω λίγο, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι τον Καλλιλέο εδώ στο Κοινοβούλιο και όπως ξέρετε παλιά τα πράγματα ήταν διαφορετικά σχεδιασμένα ε, υπήρχε το μοντέλο του ΠΠΠ παλιά αλλάξαν τα πράγματα και επιτέλους μπορούμε να ε, στήσουμε αν θέλετε το κάποιες δομές διαχείρισης για τα προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης φτιάχτηκε μια, ένας οργανισμός παλιότερα μια agency ε, υπήρχαν θέματα με τη χρηματοδότηση επανειλημμένα εμείς είχαμε πει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ένας ακόμη οργανισμός αυτά για την ιστορική ανασκόπηση και για τους συναδέλφους που δεν ασχολούνται με το θέμα τόσο ε, τόσο πολύ χρόνο ε, Ε, το λέω αυτό για να προετοιμάσω και την Κομισιόν η οποία θα πρέπει να απαντήσει και ορισμένα πράγματα για, αυτή, την, για αυτό τον οργανισμό. Τώρα, επίσης παρακάτω λέγεται ποια είναι τα καθήκοντα της, του οργανισμού αυτού η διαπίστευση ασφάλειας μάλιστα και ενδεχομένω και η εμπορική εκμετάλλευση του Γκαλιλαίου ε, και εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά πράγματα αλλά το βασικό καθήκον είναι η διαπίστευση ασφάλειας αν δεν κάνω λάθος έτσι να μου το επιβεβαιώσει και η Κομισιόν αυτό ωραία ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν τι θα πει διαπίστευση εδώ στο σχέδιο οικονομισμού διαβάζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και συζητάμε και για την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι συνδεδεμένο, είναι δεσμευμένο συνδεδεμένο με αυτήν τη διαπίστευση. Τότε λοιπόν αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο αν θέλετε για τη διαπίστευση ή η διαπίστευση δίνεται κάπου αλλού τότε τι άλλα καθήκοντα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αυτού επόμενο θέμα δομές στο εσωτερικό του οργανισμού συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και συμφωνώ και με τον εισηγητή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει και να εκπροσωπείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον στο Διοικητικό Συμβούλιο και όσον αφορά τη στάθμιση των ψήφων το 30% το ποσοστό της Κομισιόν νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της ε, Κομισιόν η οποία Κομισιόν βεβαίως ε, θα δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, ούτως ή άλλως θα το κάνει αυτό η Κομισιόν νομίζω λοιπόν ότι το 30 Νομίζω λοιπόν το 30% που προτείνει ο εισηγητής είναι επαρκές ποσοστό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να κλείνω κύριε Πρόεδρε ε, να ζητήσω άλλη μια φορά από την Κομισιόν να μας πει μερικά παραπάνω πράγματα για τον οργανισμό αυτόν τους ώστε να διασκεδαστούν και οι τελευταίες ανησυχίες και αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν σχετικά με αυτό τον καινούριο οργανισμό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, δοθούν οι διευκρινήσεις αυτές όχι μόνο επειδή με ενδιαφέρει εμένα αλλά και για να πιστούν και οι συνάδελφοι του προϋπολογισμού οι οποίοι δικαίως λένε ότι δεν θα πρέπει με το παραμικρό να φτιάχνονται καινούργιοι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος τρεις ακόμη ομιλητές Χόρν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάσον για την τόσο ενημερωτική και συνεργατική ε, προσέγγιση του. Όπως είπε και η κυρία Νίμπλε, ο Γκαλιλαίο είχε μια τριπλή ιστορία. Δεν ήταν ούτως ή άλλως μια εύκολη διαδικασία. Και πιστεύω ότι στο παρελθόν υπέφερε σαν project επειδή Ήτανε, ε, ήτανε λίγα τα κράτη-μέλη, ήταν κάποια κράτη-μέλη τα οποία είχαν κάποια ε, project, κάποιο ενδιαφέρον για το διάστημα και αυτή η Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Διαστήματος δεν ήταν κοινοτική, είχε πιο πολύ εθνικό χαρακτήρα. Και τώρα όντως ε, καλό θα είναι η Κομισιόν να διατηρήσει κάποιο έλεγχο έτσι ώστε να είναι ε, μια, ε, να έχουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό διαστήματος αυτό καθεαυτό. Γιατί όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να εποφελούνται. Ε, ίσως προχωράμε πολύ γρήγορα να πούμε 50% αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να έχουμε ένα 40% έτσι ώστε να μην στηριζόμαστε σε κάποιο κράτος μέλος, γιατί πολλές φορές μπορεί να ε, μπλοκάρουν την ψηφοφορία δημιουργώντας κάποιες συμμαχίες. Ε, ακούστηκαν σχόλια για τη ροή των πληροφοριών και οφείλω να ομολογήσω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για την έλλειψη των πληροφοριών ε, με την κυρία Νίμπλε ε, πήγαμε σε κάποιες συναντήσεις ε, για τον Γαλιλαίο που είχαμε με την Κομισιόν και το, και το Συμβούλιο και πραγματικά εξεπλάγει διότι δεν είχαμε καμία ε, ενημέρωση εκ των προτέρων. Όταν πήγαμε στη συνεδρίαση μας έδωσαν ε, διάφορες ε, πληροφορίες, ιδιαίτερα τεχνικές. Ήταν και δυσάρεστα τα νέα όσον αφορά την πρόοδο του project και είμαστε τελείως απροετοίμαστες. Γι' αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια σωστή ροή πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να χαράξουμε μία γραμμή ανάμεσα σε αυτά που προτείνει το Συμβούλιο και αυτά τα οποία προτείνει ο εισηγητής. Το Συμβούλιο δεν θέλει πουθενά να εμφανίζονται βουλευτές, διότι λένε ότι επηρεάζει την διαδικασία υιοθέτηση του προπολογισμού και ο εισηγητής θα ήθελε να έχουμε κάποιο μέλος με δικαίωμα ψήφου. Όχι όμως σαν ε, ένας βουλευτής, αλλά κάποιον τον οποίο να προτείνει το Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα για να βάλουμε σωστά, σε μια σωστή προτεραιότητα τις πληροφορίες που παίρνει το Κοινοβούλιο είναι να έχουμε κάποια μέλη, κάποιους βουλευτές, όπως είπε ο εισηγητής, ε, και αυτοί οι παρατηρητές να είναι βουλευτές όχι με δικαίωμα ψήφου, σαν παρατηρητές. Δηλαδή να ενημερωνόμεθα μεν, αλλά χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη θέση μας ε, σαν δημοσιονομική αρχή. Τώρα, το θέμα βέβαια του προπολογισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι εκτιμήσεις είναι ότι λαμβάνοντας ακόμα υπόψη και το ε, εισόδημα και τα έσοδα από τον ε, ε, από το Γαλιλαίο 550 εκατομμύρια το χρόνο εκατομμύρια το ευρώ τον χρόνο για μια απροσδιόριστη περίοδο είναι ένα τεράστιο ποσό επομένως το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι παρόντα και να μας ενημερώνουν, να μην περιμένουν να μας ενημερώνει κάποιος άλλος, κάποιος ξένος ή κάθε έξι μήνες να πηγαίνουμε σε μια συνάντηση και να μας δίνουν πληροφορίες που πρέπει να αναλύουμε μέσα σε πέντε λεπτά. Να έχουμε σωστή ενημέρωση και να ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία. Αυτά είναι τα δύο, δύο δηλαδή 40% για την Κομισιόν και δύο παρατηρητές βουλευτές στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο Εξαιρετική η έκθεση αυτή. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια θα πρέπει να περάσουμε στο 40% γιατί είμαι σίγουρος ότι με 27 κράτη-μέλη ή 30 σε λίγο θα βρίσκουμε κάποιες, κάποιους τρόπους να διαμορφώνεται μια πλειοψηφία. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι δευτερεύουν. Συμφωνώ απόλυτα με την, με την έκθεση. Συγχαίρω και τον ε, κύριο Τοσενόφσκι, τον εισηγητή. Θα ήθελα να ζητήσω μία διευκρίνηση να κάνω μία πρόταση. 30% των ψήφων στην Κομισιόν με ικανοποιεί, όμως τίθεται το θέμα της διακυβέρνησης της, της ευρωπαϊκής πολιτικής διαστήματος, όλο αυτού του τομέα. Αυτός ο τομέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποκτά τεράστιες διαστάσεις λόγω ακριβώς των όσων ε, διαβιβάζουμε, ε, ε, των όσων αποφασίζουμε. Υπάρχει ένας διευθυντής στην υπηρεσία στην του κύριου Φερχόγγιν και διαρωτώ με αυτή η διεύθυνση μήπως πρέπει να γίνει γενική διεύθυνση διότι οι συνέπειες της ε, πολιτικής του διαστήματος αυτή τη στιγμή είναι εγκάρσιες. Δηλαδή αφορούν την ανάπτυξη, τη γεωργία, την οικολογία, το περιβάλλον, δηλαδή επηρεάζουν και άλλους τομείς. Γι' αυτό διερωτώ με μήπως θα ήταν σκόπιμο το σύνολο αυτών των ε, θεμάτων ε, ε, να ληφθούν υπόψη μας και γιατί ούτως ή άλλως τα θέματα βιομηχανίας είναι σημαντικά αλλά όχι καθοριστική σημασίας. Γι' αυτό διερωτώ μήπως σε, αυτή την, σε επίπεδο διεύθυνσης μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ, ο κύριος Πάσκα. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να φροντίσουμε το ώστε η διαδρομή του Γαλιλαίου να συνεχιστεί, να είμαστε θετικοί, επικοδομητικοί, να μπορέσουμε να συσπηρωθούμε, να υπάρξει συνήθεια από όλα τα θεσμικά όργανα με την ευκαιρία επίσης θα πρέπει να πούμε μπράβο στον κύριο Τωσινόφσκι τον εισηγητή μας. Έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του, ούτω ώστε να μπορέσει να πετύχει τους στόχους μας. Θα πρέπει εμείς να ακουστεί δυνατά η φωνή του Κοινοβουλίου στην υπόθεση αυτή. Γιατί δεν είναι και λίγα τα χρήματα τα οποία ε, έχουν πέσει για αυτή την προσπάθεια. Άρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει και αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι θα πιάσουν από αυτά τα χρήματα. Άρα, συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, προσπαθειές μας τον ίδιο ρυθμό και στο μέλλον. Ευχαριστούμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριος Μπελούτσι. κλείσει την, ε, τον κατάλογο των ομιλητών. Λαμπέρ. Κύριε Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Λαμπέρ. Θα, πάρω το προ... θα ξεκινήσω με το πρώτο θέμα που είναι το πιο ευαίσθητο που είναι το δικαιώματα ψήφου της Κομισιόν στο επίπεδο του οργανισμού. Εάν η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο διαχείρισης του project, των project μάλλον, θα πρέπει να τα, μπορεί να τα διαχειρίζεται με όλα τα μέσα που θα μπορούσε να έχει στη διάθεσή της. Αντιμετωπίζουμε όλο ένα και αυξανόμενες ε, δυσκολίες με όλους τους υπολείπους οργανισμούς όπου η Κομισιόν δεν έχει ούτε δικαίωμα αρνησή ε, σε θέματα κλειδιά όπως είναι το πρόγραμμα εργασίας ή το business plan ή τον προπολογισμό ή τον διορισμό του διευθυντή. Επομένως, εδώ δεν μπορούμε να επαναλάβουμε και στην ΕΣΑ, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το ίδιο πράγμα. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε μια δυνατότητα διαχείρισης άμεση και ταχύτατη. Γι' αυτό θα πρέπει η αρμοδιότητα να βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν της ίδιας. Δεν θέλω να προβάλλω διάφορα επιχειρήματα για το 50, 30, 40 κτλ. αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε να παίζουμε την κολοκυθιά και να ε, μην παίρνουμε μια σοβαρή απόφαση για θέματα που είναι τόσο σημαντικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε την δυνατότητα να ξαναδούμε το 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν προφανώς θέλει να είναι παρόντα, είτε μέλη τα οποία εσείς τα ορίζετε, είτε με, είτε με την ε, εκπροσώπηση της ε, Επιτροπής, της Επιτροπής σας. Είμαστε στη διάθεσή σας βέβαια και να σας ενημερώνουμε άμεσα. Τώρα, ή μπορεί να είναι τα μέλη παρόντα όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις ή να είναι παρόντα και στις συζητήσεις ε, που θα προηγηθούν. Τώρα, όσον αφορά την υιοθέτηση του κανονισμού αυτού, προφανώς εμείς θέλουμε να γίνει υιοθέτηση με την πρώτη ανάγνωση. Γιατί θεωρούμε ότι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να προχωρήσουμε. Το 2010 είναι μπροστά μας. Θα πρέπει η όλη υπόθεση Γκαλιλαίο να σταθεροποιηθεί διότι ξέρουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν. Τώρα, επανέρχομαι στην παρατήρηση της κυρίας Νίμπλε. Όντως γνωρίζουμε την ιστορία, την παλιά ιστορία του Γαλιλαίου, την οποία ούτως ή άλλως εξέτασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή το ηλεκτρικό συνέδριο. Τώρα όμως ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να ευθυγραμμιστούμε με, τους, με τον κανονισμό που αποτελεί την νομική βάση. Εσείς ε, υιοθετήσατε τον κανονισμό που αποτελεί την νομική βάση. Ε, και ξέρετε τον κανονισμό ακριβώς. Θα πρέπει τώρα όμως να περάσουμε στην εφαρμογή του κανονισμού. Όλα αυτά να συγκεκριμενοποιηθούν. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Στο τέλος του 2008 ο οργανισμός έζησε έναν περιορισμό του προσωπικού της. Ο προϋπολογισμός μειώθηκε και υιοθετήθηκαν όμως και νέα καθήκοντα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε. Επομένως, Ούτως ή άλλως ο οργανισμός αυτός έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο καθορισμένο που ε, τον, τον πλαισιώνει η νομική βάση και πρέπει να περάσουμε τώρα στην ε, δράση. Δεν τελειώσατε, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, κάποιος από εσά έκανε ένα σχόλιο για το κατά πόσον θα πρέπει να δώσουμε στην Κομισιόν το δικαίωμα ε, δικαίωμα, στο δικαίωμα ψήφου γύρω στο 40%. Επαναλαμβάνω, δεν θα ε, κολλήσουμε σε αυτό το ποσοστό. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά την, ε, τα διάφορα project τα διάφορα προγράμματα τα οποία υποβάλλουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια ακόμη, κύριος Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να μιλήσω πριν το γιατί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα ήθελα, αλλά δεν ήμουν εδώ. Οπότε τώρα, ε, ρισκάροντας να παρεξηγεί ο ρόλος μου, θα ήθελα να πω τα εξής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτή τη μορφή τη διαχείριση σε σχέση με αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί για το, για το 6 ότι εμπιστοσύνη και έλεγχο χρειάζεται και όχι έλεγχο και εκ των υστέρων χτίσιμο εμπιστοσύνη. Αν θέλουμε να ε, μπορούμε να, να, να είμαστε υπεύθυνοι για το όργανο, για τη διαχείριση, θα πρέπει να είμαστε ικανοί να κάνουμε και τη διαχείριση και τον έλεγχο. Και τώρα που ρίχνω μια ματιά σε αυτή την τροπολογία που υπάρχει στο τέλο πρόταση, αναφέρει ότι σε τακτά διαστήματα θα μα ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αν ήμουν επιτροπή, τι θα έλεγα. Έχετε του δικού σα στο Συμβούλιο, στο σας Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να σας λέω εγώ τίποτα. Οπότε θα προτιμούσα να έχουμε εδώ πέρα μια διαίρεση των εργασιών και αρμοδιοτήτων ε, αυτή να ελέγχουμε τους εκτελεστικούς που θα είναι εκείνοι και εάν πάει κάτι στραβά θα, θα τους κυνηγήσουμε. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νίμπλε. Θέλει πάλι το λόγο. Ναι πρόεδρε στρέφομαι στην Κομισιόν είχα ζητήσει να μου δώσει κάποιες διευκρινίες να μου πει τι σημαίνει διαπίστευση ασφάλειας και πώς θα γίνεται αυτή γιατί όπως είπα και προηγουμένως ε, τα καθήκοντα αυτού του οργανισμού δεν είναι πολλά και θέλω να ε, δω ποιες είναι οι προτεραιότητες μπορεί η Κομισιόν να απαντήσει ρωτάει ο Πρόεδρος ε, Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο ή να απαντήσουμε αμέσως στην κυρία ή να απαντήσουμε γραπτά Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συναδελφά μου την κυρία Καβάντα για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τώρα, όσον αφορά τα καθήκοντα του οργανισμού, επαναλαμβάνω εν συντομή αυτά που σας εξήγησε ο κύριος Μπονούτσι. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού GNSS, ο οργανισμός θα πρέπει να ασκεί συγκεκριμένα καθήκοντα. Το ένα είναι η διαπίστευση, το δεύτερο είναι η εκμετάλλευση του Κέντρου Ασφάλειας Γαλιλαίων και τρίτον, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως όσον αφορά την φάση εκμετάλλευσης, που θα έρθει σε λίγα χρόνια, θα πρέπει να προετοιμάσει μέσω μελετών την, ε, την εμπορική κυκλοφορία αυτών των ε, προγραμμάτων, του Έγνος και του Γαλιλαίου πέραν αυτών των συγκεκριμένων καθηκόντων που αναφέρονται στον κανονισμό, ο οργανισμός μπορεί να έχει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει η Κομισιό μέσω συγκεκριμένης ανάθεσης. Δηλαδή το καθήκον της διαπίστευσης του συστήματος ε, είναι πολύ ευγενές καθήκον, πάρα πολύ σημαντικό και τα, ε, όσον αφορά τις δαπάνες και τα έξοδα, η πρόταση της Κομισιόν στο δημοσιονομικό δελτίο εξηγεί ποιες είναι οι ανάγκες όσον αφορά το συμπληρωματικό προσωπικό που συνεπάγεται αυτή η αρμοδιότητα. Για τα υπόλοιπα καθήκοντα, όπως σας είπε, όπως ξέρετε, είναι τα στάνταρα έξοδα, τα οποία εγγράφονται στον κανονισμό της Κομισιό, για τον οργανισμό αυτό. Σε περίπτωση που η κυρία Νίβλερ θα ήθελε να ξέρει συμπληρωματικές, να έχει συμπληρωματικές και συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες δεν έχω μαζί μου σήμερα, είμαστε στη διάθεσή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 9 ε, Δεκεμβρίου ημερομηνία κατάθεσης των τροπολογιών και μετά συνεχίζουν το 2010. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό νομίζω. Προχωρούμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης. Ο εισηγητής κύριος Γκλάντε έχει το λόγο και θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να έχετε να, μια ματιά, να ρίχνετε μια ματιά στο ρολόι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω πολλά πράγματα έτσι κι αλλιώς φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι ε, ξέρουν ε, λιγάκι το ζήτημα ή τους επισκέφθηκε ο σκιώδης ε, εισηγητής. Ε, ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε λοιπόν σε λεπτομέρειες. Εδώ το, μέχρι τώρα το πρόγραμμα ιοσκόπηση του GMES ήταν σε ερευνητικό στάδιο. Τώρα εφαρμόζεται. Πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται. Και βεβαίως ε, έγιναν πολλές σχετικές συζητήσεις πολλές φορές βέβαια ε, ερώτημα ποια είναι η σχέση με την κλιματική αλλαγή πως μπορούμε να μετρήσουμε την κλιματική αλλαγή τι μετρήσει μπορούν να κάνουν τα δορυφορικά συστήματα οι δορυφόροι που έχουμε από πιο ύψος ε, τι ακριβώς βλέπουν οι δορυφόροι ε, και βεβαίω η απαντήση είναι ότι βεβαίω όλα αυτά τα πράγματα είναι παρατηρήσιμα αν θέλετε διότι βλέπει κανείς με την αύξηση της θερμοκρασίας να μειώνονται οι όγκοι των πάγων κλπ. Από εκεί και πέρα στην Κίνα βλέπουμε να ε, ε, ε, ε να αλλάζει η μορφολογία του εδάφους αλλά αυτό δεν ε, είναι μονάχα το το το, αντικείμενο της παρατήρησης της γης δεν είναι μονάχα η παρατήρηση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής ε, με το σεισμό ας πούμε γίνεται σεισμός κάπου οι δορυφόροι μπορούν να μας βοηθήσουν ε, σχετικά με το τι έγινε με τις πλημμύρες το ίδιο ποιες περιοχές πλημμύρισαν ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο και ε, Ε, χαρτογράφηση ή άλλη δυνατότητα που θα αποκτήσουμε μέσω αυτού του συστήματος είναι η καλύτερη ε, χαρτογράφηση ορισμένων περιοχών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσο και αν σας φαίνεται περίεργο και στην Αφρική και ε, αλλού δεν υπάρχει καλή χαρτογράφηση σε κάποιες περιοχές που χρειάζεται όμως για τις επενδύσεις υποδομών κλπ. Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω τώρα για, και δεν θα αναφέρω συγκεκριμένο όνομα γιατί δεν το θυμάμαι στην νότιο-ανατολική Ασία ε, ένα παρθένο δάσος υλοτομήθηκε από κάποιους ε, και αυτό είχε ε, αναφερθεί στις ειδήσει. Ε, ωστόσο είδαμε ε, από τις ε, φωτογραφίες των δορυφόρων ότι οι υλοτόμοι αυτοί οι παράνομοι είχαν πάει στη διπλανή χώρα και είχαν για να μαζέψουν ξυλία. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το βλέπαμε διαφορετικά. Είναι χρήσιμη λοιπόν η γεωσκόπηση, η παρατήρηση της γης με δορυφόρους, ε, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχει βεβαίως όπως φαντάζεστε ε, πρόβλημα με ορισμένα στοιχεία της χρηματοδότησης ε, με διότι ο εξοπλισμός ε, και το υλικό που χρειάζεται δεν είναι ε, φθηνό όπως φαντάζεστε και βέβαια από την άλλη μεριά δεν πρόκειται να φθηνίνει αν τα αφήσει για αργότερα και αναβάλει κανείς στην αγορά ορισμένων κάποιου υλικού άρα καλύτερο είναι να αγοραστούν από τώρα ο εξοπλισμός και τελικά γιατί δεν πρόκειται να φθηνίνουν στο μέλλον ε, επίσης θέσεις ε, έχει συζητηθεί και το θέμα αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν δημοσιονομικές προοπτικές βεβαίως που πάνε μέχρι το 2013 αλλά δεν μπορούμε νομίζω να φανταστούμε ότι το 2014 το, την Άνοιξη θα παγώσουν τα πάντα διότι δεν έχει εξασφαλιστεί ε, χρηματοδότηση άρα ε, και για την προστασία λοιπόν των θέσεων εργασία πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα για τα δεδομένα τα οποία θα εισελεχθούν αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους δωρεάν ε, και βεβαίως ε, θα πρέπει να μπορεί να γίνεται ανταλλαγή των δεδομένων αυτών δηλαδή και από τις άλλες πηγές συλλογή στοιχείων θα θέλαμε να μας δίνουν δωρεάν τα στοιχεία τα οποία μπορούμε και εμείς να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε γίνεται και λόγος επίσης την ε, έκθεση εδώ και για την αξιολόγηση ε, οποία αξιολόγηση όμως θα πρέπει να γίνει αρκετά προσεκτικά διότι δεν θέλουμε να γίνουν ούτε ούτε εκεί ε, ούτε στη συλλογή στοιχείων ούτε στην αξιολόγηση ε, των προγραμμάτων και στην επεξεργασία των στοιχείων θέλουμε να υπάρχει επικάλυψη ότι υπάρχουν οι εθνικές ε, εταιρείε χαρτογράφηση σε όλες τις χώρες κλπ, κλπ που ασχολούνται με τη συλλογή στοιχείων ε, παραπέρα για τα θέματα τα πιο ε, αν θέλετε ε, γραφειοκρατικά να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που γλιτώσαμε την, ε, το βάρος της επιτροπολογίας νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα δίχως επιτροπολογία να προχωρήσουμε και βεβαίως ε, με η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ε, είμαι υπέρ της διαφάνειας ε, πιστεύω πιστεύουμε ότι μπορεί να ανατεθεί το τεχνικό αυτό μέρος στην ΕΣΑ δεν έχουμε πρόβλημα από αυτού τώρα τροπολογίες υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οφείλω να πω ε, συζητήσαμε τις συζητήσαμε Ε, μάθαμε πολλά πράγματα ίσως θα πρέπει να υποβληθεί ακόμη μια τροπολογία για την αποφυγή επικάλυψης και διπλής δουλειάς στο θέμα της συλλογής ε, στοιχείων και επεξεργασίας αυτών ε, Τώρα διαδικαστικά φαντάζομαι ότι τον Ιούνιο-Ιούλιο της επόμενης χρονιάς θα ψηφιστεί το ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω βεβαίως πώς θα λειτουργήσει το Συμβούλιο. Ε, ελπίζουμε πάντως να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα τους ώστε να μπορέσει να αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός. Ε, και κάποιο είπε προηγουμένω ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δημιουργήσει μια γενική διεύθυνση space ενδεχομένω διάστημα, δεν ξέρω πώ θα λέγεται. Είναι γεγονό ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με το διάστημα. Δεν ξέρω, δεν είμαι αντίθετο στην ιδέα, αλλά θα δούμε. πρόεδρο. ωραία, έχω τέσσερι ομιλητέ άλλο που θα το λόγο, παρακαλώ. Lamberts. Okay. Just in time. <laughs> Ähm, dann darf Θα ήθελα να ξεκινήσω τον κύριο Ρεμέκ. Ε, děkuji, Já co a e, co z nás Πρόεδρε, τι, δεν μιλάνε τίποτα. Τα περισσότερα έχουν αναφερθεί. Μην τα επαναλάβω, αλλά να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο το οποίο επετέλεσε. Επίσης, ε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με το κείμενό του και θα ήθελα να σταθώ σε δύο τροπολογίες που τις χωρίασε και ο εισηγητής πρώτα πρώτα όσον αφορά την συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών πρώτα πρώτα και ε, θα πρέπει να προσέξουμε σχετικά με αυτό την ε, μεταβατική περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει τους ε, αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Δεν κατάλαβα το όνομά μου μάλλον, πρόεδρε, όταν μου δώσετε το λόγο. Συμπαθάτε με, λέει ο Έχω να σας πω τα εξή όσον αφορά το λόγο πρόγραμμα. Πρώτα-πρώτα. Πρόκειται για το κατά πόσο θα συνεχιστεί υπάρχει το υπηρεσμό το 2013 σχέση με την μακρά διάρκεια του προγράμματος και επίσης σε σχέση με την πρικοδότησή του. Έχουμε 150 ευρώ τα οποία που καταρχήν προβλέπονται αλλά δεν αρκούν. δεν προβλέπεται κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση των, ε, των, των, των εκτοξεύσεων των δορυφών. Άρα θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Τώρα, όσον αφορά τα δεδομένα, συμφωνώ με την ε, ανοιχτή πρόσβαση, όπως πρότεινε ο εισηγητή, γιατί στόχος του προγράμματος βασικός είναι το να ξεκινήσει μια τέτοια αγορά ε, επί τη βάση αυτών των raw data όπως θα βγαίνουν από το πρόγραμμα. Και βέβαια στα πλαίσια αυτού του προγράμματος θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και την καινοτομία. Όλες οι σχετιζόμενες των το GMS e δεν έχουν ακόμα περιχαρακωθεί, δεν έχουν οριστεί, οπότε προσοχή όσον αφορά το κατά πόσο πρόσβαση θα είναι ελεύθερη ε, και πώς αυτό θα κατοχυρωθεί από την νομοθεσία. Επίσης να δούμε πώς θα υπάρχει η ασφάλεια για τις ε, ε, πληροφορίες, πώς θα εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών και πώς θα προστατευτούν οι χρήστες αυτών των πληροφοριών. Τώρα για την κυριότητα και ρόλο των operators όσον αφορά την υποδομή. Θα πρέπει να βρούμε το πιο αποτελεσματικό σχήμα που να αποδίδει. Μια που από ένα σημείο και μετά θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση της ε, υποδομής. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βαλιάν, ναι, έτσι, έτσι δεν λέει το Ναι, ναι, ναι, έτσι. Τσίτσεστερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ, όπως οι άλλοι συνάδελφοι, να συγχωρώ τον κύριο Γκλάντε. Ε, σε ένα σημείο μόνο διαφωνώ όπως είπε, αλλά θα ήθελα να υποβάλω και κάποιες προτάσεις και τρεις-τέσσερις ε, τροπολογίες τις οποίες θα προτείνω επίσης. Όσον αφορά την επικάλυψη των πληροφοριών, θεωρώ ότι είναι πιθανό η συλλογή νέων πληροφοριών να οδηγήσει σε επανάληψη και επικάλυψη σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. και ότι αυτό να μην αποτελέσει φραγμό στη λειτουργία του GMS. E Δεν νομίζω αυτό το σημείο το καλύπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ε, πρότασή της. Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι αυτό το πρόγραμμα Προποθέτει να εμπλακούν μία σειρά ενδιαφερομένων. Ελπίζω ότι αυτό θα ληφθεί υπόψη και θα εξασφαλιστεί όσο γίνεται ευρύτερη διαβούλευση. Τώρα το τρίτο και τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω, ε, σημείο το οποίο διαφωνούμε με τον ε, εισηγητή και τον έφερε κύριε Βαλιάν είναι η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες του GMS εγώ σας προτείνω και υποβάλλω την επιφύλαξή μου διότι είπαμε ότι δεν προβλέπεται ικανή πρικοδότηση και άρα το να είναι ελεύθερη πρόσβαση μου φαίνεται λίγο βιαστική η ρύθμιση. Όσον αφορά τώρα την ε, συγκρότηση μιας αγοράς για αυτές τις υπηρεσίες δεν ξέρω αν αυτό θα πιάσει τόπο αυτή η προσπάθεια αν είναι δωρεάν η παροχή των υπηρεσιών και ποιο θα, κάνει κάτι, θα κάτσει να ενδιαφερθεί για κάτι το οποίο δεν θα αποδίδει κάποιο κέρδος. Άρα έχω την επιφυλαξή μου και παρακαλώ να η υπόψη. Καταλαβαίνετε ότι έχει τις ε, θέσεις του ο κύριος Γκλάντερ κάποια στιγμή ίσως ε, συζητηθεί περισσότερο. Η κυρία Τατή. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπλάνκ για το σχέδιο έκθεσης το οποίο μας παρουσίασε σήμερα. Είναι αλήθεια ότι σαν σκιώδης εισηγητήρια του ΕΛΚΑ δεν έχω να κάνω ουσιαστικά σχόλια για αυτό το σχέδιο. Απλώς κάποιες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω για την πρόταση κανονισμού και το σχέδιο έκθεσης. Μία, μία, για μια τροπολογία που αφορά την συνέχεια των δεδομένων που είναι και η εγγραφή στον κανονισμό της ε, διατήρησης των στοιχείων και της συνέχεια των δεδομένων, δηλαδή να είναι ε, συνεχώς προσβάσιμα. Δηλαδή θα πρέπει να μπορούν οι χρήστες να χρησιμοποιούν με πλήρη εμπιστοσύνη το σύστημα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και το, την πρόταση αυτή να την εντάξουμε στο κείμενο αυτό καθε και όχι στα, στην ιδεολογική σκέψη. Γιατί δεν έχει την ίδια νομική ισχύ, δεν τονίζει αυτή την αρχή της συνέχειας των δεδομένων. Δεύτερον, όσον αφορά την χρηματοδότηση. Αυτό, που, αυτό που ελέγχθη Ε, προσπαθώ να τα πω σωστά τα ονόματα, αλλά δεν τα λέω καθόλου. Ε, για ε, το θέμα της χρηματοδότησης εθίχθη. Εγώ νομίζω, το είπαμε και στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε τον Οκτώβριο, ότι εδώ υπάρχει μία έλλειψη διαφάνειας στην χρηματοδότηση και στον κανονισμό. Πιστεύω ότι ο κανονισμός οργανώνει κάποια πράγματα και όμως η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι καλύτερα οργανωμένη και καλύτερα και να παρουσιάζεται καλύτερα έτσι ώστε να έχουμε και μια ισορροπημένη παρουσία των υπηρεσιών. Έτσι όπως έχει το πράγμα τώρα δεν υπάρχει σωστή επίβλεψη του θαλάσσιου χώρου ε, και του ενέργειου χώρου. Θα πρέπει οι τέσσερις ε, υπηρεσίε γεωσκόπησης ε, να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο οριμότητας. Αυτό δεν φαίνεται στο κείμενο. Επομένως θα πρέπει ο κανονισμός ε, καταρχάς ε, να αντικατοπτρίζει την ισότητα, την δημοσιονομική ισότητα όλων των υπηρεσιών. Τώρα, ε, δικαίωμα πρόσβαση στις, ε, στα δεδομένα. Ε, Κάποιο συνάδελφος προηγουμένω αναφέρθηκε στο αν είναι δωρεάν η πρόσβαση ή θα πρέπει να πληρώνουμε κτλ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση που σχετίζεται με τροπολογία 3 και 12. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την αρχή του δικαιώματο πρόσβαση. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε δικαίωμα στην πρόσβαση και από εκεί πέρα, αν είναι δωρεάν ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένε πληροφορίε που δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους, ακόμα και αν είναι επιπληρωμή. θα μπορούσε το GMS να είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και των, και πολιτών ΜΕΝΑ, αλλά θα πρέπει να δούμε ε, αυτοί οι περιορισμοί που προτείνουμε, τι κόστος ε, θα συνεπάγεται, γιατί όταν οι περιορισμοί κοστίζουν. Τώρα, μία τροπολογία, στο, η τροπολογία 8 μάλλον, ε, θα εγγυάται την ε, ακαιρεότητα των δεδομένων ε, του ΖΕΜΕΣ. είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την διαπίστευση των δεδομένων και την πιστοποίηση μάλλον των δεδομένων για να μπορέσουμε να έχουμε μία χρήση των δεδομένων αυτών μέσα στα πλαίσια της ρύθμισης των κρίσεων και των προβλημάτων. Παραδείγματος χάρη όταν έχουμε κάνει με οικολογικές καταστροφές. Ένα άλλο θέμα είναι η διακυβέρνηση το οποίο το συζητήσαμε νομίζω. Υπάρχει μια έλλειψη διαφάνειας, παρά το ότι ξέρουμε ότι η καλύτερη διακυβέρνηση είναι υψής της σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος αυτού. Ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα ε, θεσμικά όργανα της κοινότητας. Ε, η, στις 12 του μηνός η, Νοεμβρίου η Κομισιό κάνει, έχει κάνει μια ανακοίνωση που όμως δεν καθορίζει λεπτομερώς και συγκεκριμένα τις διάφορες αρμοδιότητες ε, αρμοδιότητες ε, που έχουν οι διάφοροι φορείς του και εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του καθένα και θα πρέπει εκτός από τη διαχείριση των χρημάτων να υπάρχει και διαχείριση των δομών. Δηλαδή τα εθνικά κράτη-μέλη και, οι και τα θεσμικά και τα κοινοτικά όργανα διαχειρίζονται τις, ε, τις υποδομές και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πιο αποτελεσματικό, ε, μια πιο αποτελεσματική διαχείριση και των υποδομών και των κονδυλίων. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία για μας και δεν θα πρέπει να τη χάσουμε. Ευχαριστώ. Uh, uh, Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γκλάντε για την εκθεσή του. Κύριε εάν δεν συναντηθήκαμε νωρίτερα, ε, ε, αυτό οφειλότανε στο ότι δεν χρειαζόταν να έρθω να σας βρω. Σε, σε αυτό που είπε η κυρία Τατή, ότι η πρόσβαση για Ευρωπαίους και άλλους προβλέπεται και αυτό επί τη βάση της αμοιβαιότητας. Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, είναι πολύ σπουδαία υπόθεση αυτό το πρόγραμμα και δεν γίνεται να έχουμε παγκόσμια κάλυψη από πλευρά παρατήρηση αν οι ενδιαφερόμενοι δεν κάνει ο καθένα αυτό που πρέπει. Ινδία, Βραζιλία, η Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία. Ε, εάν αυτοί κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, τότε, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Ε, όμως, είναι πάρα πολύ σημαντική η αμοιβαιότητα, τουλάχιστον όσον αφορά κάποιε χώρε, κάποιε φορεί που μπορούν, έχουν δυνατότητα να κάνουν το ίδιο. Γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Να κάνουμε εμεί τη δουλειά των άλλων και υπάρχουν και άλλε χώρε που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, αλλά όμω ε, μιλάμε τώρα για άλλη ρυθμίση. Άρα θα πρέπει να γίνει σαφής ε, διάκριση μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Τώρα θα ήθελα να συμφωνήσω στον αφορά την ελεύθερη προσβασιμότητα. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ ακριβό και δεν ε, διανούμεθα να το ξεκινήσουμε και μετά να, ε, να το, το εγκαταλείψουμε. Ξέρουμε, προς τα πράγματα ξέρουμε τι στρατηγική θα χρειαστεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε και όπως είπες και εσύ, Τσόλς, θα να δούμε μήπως ευθύς εξ αρχή έχουμε μία ελληπική χρηματοδότηση. Και αυτοί που θα χρησιμοποιούν το GMS για μη κερδοσκοπικούς λόγους, αυτοί όντως να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόταση όμως κάποιες εταιρείε που θα βγάλουν κάποιο θεμητό κέρδος από αυτά τα, τα μη στοιχεία του GMS ε, πιστεύω ότι αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να κάτι να δίνουν από αυτά τα οποία ε, τους, τους, τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, προσοχή να μην υπάρξει διακινδύνευση. Μην ρισκάρουμε όλη την υπόθεση, γιατί έτσι μπορεί κάποια στιγμή να μην υπάρχουν τα χρήματα να, να συνεχίσει να τρέχει το πρόγραμμα. Τσάρλ. έχεις δίκιο και θα σε βοηθήσω με τροπολογία που μπορώ, θα προτείνω. Βέβαια. Με πάρα πολύ σύντομα να σας πω σε σχέση με την πρόσβαση ήδη είχα τοποθετηθεί συνεργασία με την κυρία Ντατή πριν από καμιά κάνα δίμηνο νομίζω και συμφωνώ 100% με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γκλάντα και το κείμενό του μας λέει να υπάρχουν υπηρεσίες για όλους τους ε, Ευρωπαίους και έτσι να αναπτυχθεί μια ολόκληρη αγορά, να ωφεληθούν οι ΜΜΕ. Απλώς όμως θα ήθελα να δούμε τι έγινε πρόσφατα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Εκεί έχουν τον ε, δορυφόρο Αμσάτ. Και εδώ 40 χρόνια έχουν τον δορυφόρο, οπότε τα αρχεία εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, είναι υπολογίσιμα. Ε, Βεβαίω όμω η πρόσβαση εκεί πέρα ε, γίνεται κατόπιν αντιτίμου, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ υψηλό. Και έχει 20.000 επισκέψεις και αγορά στοιχείων ανά έτος. Και τώρα έχουμε 200.000 ανά μήνα. Καταλάβετε την παραπηρημιουργία της αγοράς. Οπότε θα πρέπει και εμείς να θέλουμε να εντονώσουμε την καινοτομία να έχουμε ανάλογη εξέλιξη. Μαζική ανάπτυξη, μετά αφού συγκροτηθεί η αγορά και κατόπιν βλέπουμε πώς θα γίνει η χρηματοδότηση από αυτούς που αποκομίζουν κέρδος. Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου πρέπει να δευτερολογήσω γιατί θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντατή για τις διευκρινήσεις της βεβαίως και είναι σωστό το να έχουμε ε, την διάκριση μεταξύ ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης βεβαίως και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα. Όμως νομίζω ότι δεν θα ήταν ε, τόσο συνετό το να αποκλείσουμε τρόπους χρηματοδότησης. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας ε, για, την, ε, για το ενδιαφέρον που δείχνει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Γεωσκόπησης. Να πω ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η αρχή των δεδομένων που είναι μια αρχή στην οποία στηριχθήκαμε για να αναπτύξουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης και να επιστήσω την προσοχή σας στις συνέπειες που έχει αυτή η συνέχεια των δεδομένων και στην διατήρηση και στη μονιμότητα των δομών των διαστημικών αλλά και στην διατήρηση των υπηρεσιών, την σταθερότητα των τεχνικών αρμοδιοτήτων στην Ευρώπη αλλά και ε, την, στη δυνατότητα της χρηματοδότησης και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ανακοίνωση που υιοθέτησε η Κομισιόν στις 28 Οκτωβρίου και που αφορά στα θέματα της ε, διατήρησης ε, ε, μονιμότητας, αν θέλετε, των διαστημικών υποδομών θα πρέπει μέχρι το 2011 να έχουμε μια επαγγελματική αν θέλετε αντιμετώπιση έτσι ώστε να, ε, των υποδομών αυτών έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριος Γκλάντε. Ναι, ναι, ε, ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις που έγιναν και για τα σχόλια. Βεβαίως θα ε, φροντίσω να τα λάβω υπόψη τώρα για την επικάλυψη ε, στοιχείων, για τη συλλογή των στοιχείων κτλ. Όντως ε, κάπου θα πρέπει να το βάλουμε αυτό τώρα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. Ξέρω πώς ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα στα διάφορα κράτη-μέλη αλλά και στη δική μου χώρα ε, ε υπάρχουν διαδικασίες που εγκρίνουν την αποστολή πρώτα-πρώτα του καθενός από αυτούς τους δορυφόρους θα πρέπει να βρούμε και εκεί μια λύση που να γίνει αποδεκτή από όλους τώρα για τη χρηματοδότηση είναι σίγουρο ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε ξανά τα πράγματα αυτά αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε ένα ε, μια συνεργασία ε, σε μια πρώτη φάση δεν ε, πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς δεν, δεν πρόκειται να διαχειριστούμε αν θέλετε το όλο σύστημα σαν να ήταν επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα στο μέλλον μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και τότε θα πρέπει να συζητήσουμε αν κάποια στοιχεία θα δίνονται δωρεάν ή όχι και τα και τι θα γίνει με την εμπορική τρόπο την εκμετάλλευση του συστήματος. Ευχαριστώ λοιπόν άλλη μια φορά για τις προτάσεις και τα σχόλια. Θα κάνω κάποιες αλλαγές αλλά θα υποβάλλετε τις τροπολογίες σας αν θέλετε μέχρι το τέλος των, της προθεσμίας ε, εκείνο το οποίο περιμένω με ανυπομονησία είναι να δω τι θα γίνει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, για την κατάθεση των τροπολογιών. Ε, η προθεσμία είναι 10 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Προχωρώ στο σημείο 8 της σημερινής διάταξης για την ε, μελέτη που έγινε σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Λέων Σεράνο ο οποίος θα μας παρουσιάσει το ζήτημα αυτό και φαντάζομαι ότι θα γίνει και μεγάλη συζήτηση μετά. Λοιπόν, κύριε Σεράνο, έχετε το λόγο. Μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω πρώτα πρώτα ποιο είναι τα συμπέρασμα αυτής της έκθεσης ούτω ώστε να υπάρχουν στη συνέχεια και ε, κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις. Να δούμε πρώτα πρώτα τα θέματα της διακυβέρνησης. Είναι το θέμα μας στα πλαίσια της αξιολόγησης της, ε, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Να καταλάβουμε επίσης το ευρύτερο τοπίο. Μην μιλήσουμε δηλαδή μόνο για την, ε, για την έρευνα, αλλά και για τις πολιτικές που έχουν σχέση με τη γνώση, που είναι όλες πάρα πολύ σημαντικές. Ούτως ώστε να δούμε όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πώς εξελίσσονται. Το Κοινοβουλίο λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε τις πρωτοβουλίες του, επιβάσει του άρθρου 169 και 171 με βάση της παλαιάς αρρύθμισης των ε, άρθρων. Ξέρω ότι αυτό τώρα με τη συνθήκη καινούργια θα αλλάξει, Όμω, επίση να δούμε τι άλλε ε, πρωτοβουλίε υπάρχουν, τι άλλο, ούτω ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα εμφανιστεί μετά και θα συμπληρώσει την σημερινή μας πρωτοβουλία. Όταν μιλούμε για χώρο έρευνα, μιλούμε και για τις κοινοτικέ προσπάθειες αλλά και των κρατών μέλλον στο πλαίσιο της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα, σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε το, το πόσο η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει ένα ευρύτερο πλαίσιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Κάποιες φωτοβουλίες προέρχονται από τα κατημέλη και κάποιες από την κοινότητα. Άρα να μην θεωρούμε ότι όλε οι πρωτοβουλίε αφορούν μόνο τα κοινωτικά όργανα, αλλά και ο ρόλο των είναι πάρα πολύ σημαντικό Και λόγω τη χρηματοδότηση που γίνεται, αλλά και η ίδια η πρωτοβουλία αποτελεί πολλές φορές δέσμευση υποχρέωση των κρατών μελών. Επίση, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η, ποια είναι η διάσταση τη διακυβέρνηση από πλευράς των πρωτοβουλειών της ε, έρευνας. Και γι' αυτό μελετούμε και αυτή τη διάσταση και αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν το πώς γίνεται η διακυβέρνηση της έρευνας. Μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποιες από αυτές τις πτυχές καλύπτονται κάθε φορά την πρωτοβουλία. Ας πούμε το πόσο ανοιχτή είναι μια πρωτοβουλία. Πόσο δηλαδή μπορεί να καλύψει τα συμφέροντα των εμπλεκομένων. Η διαφάνεια. Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων. Χρήση πόρων και επικοινωνία των εμπλεκομένων. Τι σημαίνει δηλαδή στον κανονισμό, διαφάνεια και πώς εκφράζεται μετά. Ισορροπίες, ισορροπίες μεταξύ των συμφερόντων και της εκπροσώπησης των ε, εμπλεκομένων κάθε φορά. Αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρήση των πόρων σε σχέση με τους στόχους που τάσσονται κάθε φορά. Μπορεί να υπάρχουν επομένω και κάποιε πολύ μακρόπνοε πρωτοβουλίε, γιατί οι στόχοι θα πρέπει να προσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα αν όχι κάθε χρόνο και να υπάρχει προσαρμογή αυτών στο τι ενδιαφέρει του εμπλεκόμενου. προσαρμοστικότητα και ευελιξία θα πρέπει να προκύπτουν κάποια αποτελέσματα και η κοινωνία να τοποθετείται και να ανταποκρίνεται σε αυτά τα αποτελέσματα. Το timing τώρα. Ο χρονισμός, δηλαδή το, το, το πότε λαμβάνονται οι αποφάσεις, κάτι το οποίο αφορά την πρωτοβουλία και τις εσωτερικές λειτουργίες και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει συγχρονισμός όσον αφορά τι δραστηριότητε που υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Τέλο, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διεθνοποίηση. Δηλαδή, το σε, σε ποιο βαθμό σε κάποιο πρωτοβουλίο μπορεί να συμμετάσχουν και οι τρίτε χώρε. Αν ε, η, ο ερευνητικό χώρο είναι ανοιχτό στον υπόλοιπο κόσμο και πόσο εύκολο μπορεί να μετάσχουν τρίτο χώρο. Επί τη βάση όλων αυτών τώρα θέλω να δούμε κάποια συμπεράσματα, κάποιες συστάσεις που προκύπτουν. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται. Πρόκειται για ένα στοιχείο που κινητοποιεί την κοινότητα για να κάνει μεταβολές, αλλαγές στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία. Άλλο συμπέρασμα είναι ότι αυτό το Ιωνί σταθερό σενάριο αφορά ένα χώρο λιγότερο ξεκάθαρο όπου η συμμετοχή δεν είναι τόσο αυστηρά καθορισμένη. Προσπαθούμε εδώ πέρα να βρούμε καινούριου τρόπους, ούτω ώστε να έχουμε μια διακυβέρνηση που να καλύπτει τις πρωτοβουλίες της ΕΡΑ, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. Θα πρέπει να δούμε επίση το, το υψηλό κόστο που έχει σχέση με την υλοποίηση των πρωτοβουλειών και τη χρήση των μέσων που έχει η ΕΡΑ. Θέλουμε όλο ένα και περισσότερε πληροφορίε να υπάρχουν όσον αφορά τη διαδικασία τη ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση. Τώρα, για την διακυβέρνηση τη ΕΡΑ. Θα πρέπει τα προβλήματα κάπως να επιληθούν, γιατί εδώ έχουμε μια σειρά πρωτοβουλειών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις της υλοποίησης των πρωτοβουλειών βάση ανάλυση που έχουμε κάνει διαπιστώσαμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ευελιξία στη διακυβέρνηση. Συνέπεια της ευελιξίας είναι ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην προσέγγιση. Κάτι το οποίο θα αυξηθεί όταν έχουμε τις νέες πρωτοβουλίες. Και θέλουμε να υπάρχει αυτή η ευελιξία και η ποικιλία στη διακυβέρνηση. Για αυτούς που συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, που μπορεί ο καθένας να βρει ένα σχήμα το οποίο μεταβάλλεται από τη μία πρωτοβουλία στην άλλη. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε την προσαρμογή όλων αυτών των ε, πρωτοβουλειών. Επίσης, να δούμε τον ρυθμό με τον οποίο προσαρμόζεται το κάθε κράτος μέλος αυτής της πρωτοβουλίας τα προγράμματα δεν συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Με αυτό αφετηρία διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιες συστάσεις δικές μας τόσο ώστε να επιταχυνθεί η δημιουργία της ΕΡΑ. Αυτό αφορά τα κρατημέλη και την προσαρμογή τους, την ευελιξία τους σε σχέση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τι επιτάχυνση μας μπορεί γίνει τη υπόθεση αυτή σε επίπεδο κράτους μέλους. Ε, το θέμα είναι εδώ το ότι δεν έχουμε το, το, το ίδιο άνοιγμα σε κάθε κράτος μέλος. Και αυτό θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα εθνικά προγράμματα. Το ίδιο ισχύει και με, την, ε, με τα κονδύλια τα οποία πάνε σε κάποιο κοινό κορβανά για τις πρωτοβουλίες της ΕΡΑ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πλαίσιο όπως το πλαίσιο του ότι προηγούνται, προηγούνται οι ανθρώπινοι πόροι και κατόπιν η οικονομική. Θα πρέπει να υπάρχει ομοιογένεια στο πλαίσιο το οποίο διέπει τις ε, πρωτοβουλίες της ΕΡΑ. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και κινητικότητα όσον αφορά τους υπάλληλους που ασχολούνται με αυτές τις πρωτοβουλίες. Και άρα θα πρέπει να αρθούν οι φραγμοί για να μπορεί να κινηθεί κάποιος και σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, είναι χρήσιμο να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την έρευνα με την ανωτάτη παιδεία. Uh, και έτσι να υπάρχει κάποιο είδου παροχή συμβουλών συγκεκριμένων για αυτές τις πολιτικές και με κάποια μόνιμα σχήματα να διευκολύνεται η συζήτηση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές. Ακόμα και στην Κομισιόν. Και έτσι να δούμε πώς οι πολιτικές της γνώσεις θα συντεριάξουν με το αέρα. Άλλες συστάσεις αφορούν το πώς θα είναι πιο ελκυστικές αυτές οι πρωτοβουλίες προς τους εμπλεκόμενους. και έτσι να έχουμε την καλύτερη συμμετοχή. Σωματεία, μικροσκοπικοί οργανισμοί εκτός Ευρώπης ε, έχουν πρόβλημα σχέση με τη συμμετοχή τους και άρα θα πρέπει να, να βαθμιστεί ο ρόλος τους. Το ίδιο ισχύει και το ίδιο προκύπτει αν αναλύσουμε τι είδους χρηματοδότηση έχουν αυτοί που συμμετέχουν. Αλλάζουν οι κανόνες συμμετοχής έτσι κι αλλιώς και άρα αλλάζει και το, ο τρόπος της χρηματοδότησης. Όμως όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλία δημιουργείται πρόβλημα. Ιδίω όταν ε, έχουμε συγχρηματοδότηση και θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα των πλαισίων που διέπουν αυτή τη χρηματοδότηση από τη συγχρηματοδότηση. Να υπάρχει κάποια συνέχεια μέσα στη ρύθμιση, κάποια συνέπεια και να μην ξεκινάμε κάθε φορά από το α. Παρακάτω πώς μπορούμε να καλύψουμε και να ελκύσουμε και μη Ευρωπαίους. Πώς δηλαδή θα ανοίξει η αίρα και για πρωτοβουλίες που απευθύνονται στον υπόλοιπο κόσμο. Να απλουστευτεί η διαδικασία, να έχουν τέτοιες παγκόσμιου χαρακτήρα πρωτοβουλίες και με μνημόνια κατανόηση να διευκολυνθούν τα πράγματα. Που θα είναι γενικού χαρακτήρα αυτά τα μνημόνια. Και να συμμετέχουν Ευρωπαίοι και μη Ευρωπαίοι. Επίσης η έκθεση προσφέρει κάποιες συστάσεις για τις πρωτοβουλίες 169 και 171 θα ήθελα απλώς να τονίσω κάποιες από αυτές, παραδείγματο χάρη διότι είναι ανάγκη να ε, επανεξετάσουμε τον τρόπο που συζητάμε τις ε, διαδικασίες έγκρισης αυτών των πρωτοβουλειών, διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, επιταχύνουμε την παρουσίαση και την έγκριση αυτών των προτάσεων, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν έναν ρόλο, σωστό ρόλο θα πρέπει να έχουμε μηχανισμούς που να ε, καθορίζουν τον τύπο των πρωτοβουλειών που θα πρέπει να υιοθετήσουμε στο μέλλον και να προσφέρουν στο Συμβούλιο κάποια στοιχεία, κάποια δυνατότητα να τα συζητήσει όλα αυτά. Εκτός από τον σημαντικό ρόλο που παίζει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή για την εξέλιξη αυτών των πρωτοβουλειών. Επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, εξασφαλίσουμε τις αλλαγές, ε, τις δομικές αλλαγές για την διακυβέρνηση. Από τη στιγμή που εγκριθούν ε, οι πρωτοβουλίες τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον για τα επόμενα 7-8 χρόνια πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης και διαχείρισης κάποιες ευελιξίες. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε ε, και κάποιες διαδικασίες ε, έτσι ώστε να επιτρέψουμε διάφορα επίπεδα δέσμευσης. Η έκθεση εξασφαλίζεται σαν, ένα, σαν ένας μηχανισμός όπου ε, διασφαλίζει την διαφάνεια, κυρίως αναφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Θα πρέπει να, ξέρουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην, ε, στην χρηματοδότηση. Και είναι απαραίτητο όλοι να γνωρίζουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Επίσης, η έκθεση αντιμετωπίζει κάποιες συγκεκριμένες ε, συστάσεις ε, για κάποιες πρωτοβουλίες που εμφανίζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο, το ERANET. Επίσης, στην έκθεση αυτή ε, αναφερόμαστε σε αυτές τις συστάσεις γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις το, ότι χρησιμοποιούν προς ε, ε, έναν μηχανισμό μετάβασης προς άλλα σχήματα του ΕΡΑΝΕΤ. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ε, πώς μπορούμε να οδηγηθούμε και σε άλλες πρωτοβουλίες, π.χ. πρωτοβουλίες του άρθρου 169. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν διάφορες συστάσεις για το άρθρο 169 και 171, αλλά και στις δύο αυτές περιπτώσεις το πιο σημαντικό μήνυμα είναι να πούμε ότι συστήνουμε δύο πράγματα για τους κανό, κοινούς κανόνες διακυβέρνησης για όλους και αυτό γιατί, διότι εάν έχουμε έναν, ένα σώμα, αν θέλετε, κοινών κανόνων και μια, κάποια ευελιξία έτσι ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες ιδιαιτερότητες, αυτοί οι κοινοί κανόνες διευκολύνουν και τη συμμετοχή ε, γιατί οι συμμετέχοντες όταν συμμετέχουν σε, κάποιο, σε κάποια πρωτοβουλία ΕΡΑΝΕΤ και αλλάξουν πρωτοβουλία πάνε σε μια άλλη πρωτοβουλία της ΕΡΑΝΕΤ θα ε, αντιμετωπίσουν τους ίδιους κανόνες θα αισθάνονται δηλαδή κάπως σε οικείο περιβάλλον το ίδιο ισχύει και με τις, ε, και με τις πρωτοβουλίες του άρθρου 171 Επίσης εξετάζουμε και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν κάποιες πρωτοβουλίες, κοινές πρωτοβουλίες τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη βελτίωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας ε, δηλαδή ε, τις, τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ε, αντιμετωπίζεται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές έρευνας, δημιουργείται ένα κονσόρτσιουμ ε, και αυτό ε, χρησιμοποιείται σαν βάση για να ξεκινήσουμε νέες υποδομές για την ε, ευρωπαϊκή έρευνα και θέλουμε να διευκολύνουμε την ευρω... τον εξευρωπαϊσμό θα έλεγα, τον εξευρωπαϊσμό αν μου επιτρέπετε τον όρο των υποδομών των εθνικών και των υπερεθνικών ε, υποδομών έρευνας. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με άλλα στοιχεία τα οποία θα βοηθούσαν τις ε, υποδομές τεχνο, τις τεχνολογικές, της έρευνας, να ενταχθούν καλύτερα στο οικοσύστημα. Θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε τους ε, μηχανικούς, τους ερευνητές, ε, μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας νέων δομών έρευνας. Και αυτό έχει ένα πλεονέκτημα διότι γνωρίζουμε στο σύνολό του τον ε, τομέα και ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εν κατακλείδη εξετάζουμε και άλλες πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Τεχνολογίας ε, και Γνώσης που θα εγκριθεί και θα ξεκινήσει στο τέλος της, του έτους και του χρόνου θα βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής. Και μετά ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βοηθήσει την προώθηση των πολιτικών γνώσης στην Ευρώπη. Δηλαδή να έχουμε με υψηλή εκπαίδευση ε, και καινοτομία και έρευνα. Ε, και Τα θέματα τα οποία καλύπτουν επίσης πάρα πολύ σημαντικά και για να μην ε, χρονοτριβήσουμε περισσότερο κάποιες τελικές παρατηρήσεις θεωρούμε ότι μια σωστή και αποτελεσματική διακυβέρνηση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας θα αποτελέσει ένα αριστούργημα και ένα, ε, τον ακρογωνίο λίθο για την επιτυχία των πολιτικών της ευρωπαϊκής έρευνας ε, ο ορισμός των κοινών κανόνων ε, φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικός ε, για να επιταχύνει και να διευκολύνει την εφαρμογή των πρωτοβουλειών της, του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας θα έχουμε κοινού κανόνε ε, που είναι κοινοί και για τις πρωτοβουλίε ε, του άρθρου 169 και του άρθρου 171. Τώρα μπορεί να έχουμε στο μέλλον ε, και άλλες πρωτοβουλίες σε συνδυασμό ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Εντάξει, μπορούμε να έχουμε κάποια συζήτηση για να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να εφαρμοστούν αυτέ οι πρωτοβουλίε. Επίση, ε, σε διεθνέ επίπεδο είπαμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνα σε όλο τον πλανήτη. Ε, θα πρέπει να έχουμε... Ε, θα πρέπει να διευκολύνουμε τις διακυβερνητικέ συμφωνίες έτσι ώστε να, επιταχύνουμε και να διευκολύνουμε την διεθνή ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα Με την παρουσίαση της μελέτης. Τρεις ζήτησαν τον λόγο μέχρι τώρα. Ο κύριος Τσουκαλάς πρώτα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή για την ωραία του έκθεση και να σας ξαναευχαριστήσω σας κύριε Πρόεδρε γιατί τον τελευταίο καιρό με ευχαρίστηση βλέπω ότι τα ζητήματα έρευνας και τεχνολογίας είναι συχνά στην ατζάντα της Επιτροπής μας, πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ ε, ευχάριστο. Η έκθεση που μας παρουσιάστηκε μιλάει για εντό εισαγωγικών difficulties observed in the attainment of the Lisbon strategy quantitative targets. Πρόκειται νομίζω για μια σημαντική υποτίμηση της πραγματικότητας και είναι ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο του στρογγυλεμένου τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε τα θέματα έρευνας και στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής δυστυχώς. Από την άλλη πλευρά ορθά περιγράφεται και επισημαίνεται η πολυπλοκότητα των διαφόρων πρωτοβουλειών που έχουν ληφθεί στα πλαίσια της ΕΑΡΑ και αυτές είναι πολλές. Πλαίσια, δομές, οργανισμοί, φορείς. Φαίνεται καθαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά διαρκώς προς ένα σύστημα αυξανόμενης πολυπλοκότητας όσον αφορά τη διαχείριση και χρηματοδότηση της έρευνας. Και αυτό είναι αυτονόητο ότι γίνεται σε βάρος της αποτελεσματικότητας. Πολύ φοβάμαι ότι αντί να χρηματοδοτούμε πειράματα, πειραματιζόμαστε με τις χρηματοδοτήσεις. Αντί να κάνουμε πολιτική έρευνα, ακόμη ερευνούμε την πολιτική μας. Και το πρόβλημα της ευρωπαϊκής έρευνας δεν είναι τελικά οι ερευνητές της, αλλά αυτοί που δημιουργούν και εφαρμόζουν πολιτική έρευνα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό όταν υπάρχουν γύρω μας παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών και πολιτικών έρευνας τόσο στον υπόλοιπο κόσμο όσο και μέσα στην Ευρώπη. Θα μπορούσα για παράδειγμα να αναφέρω το παράδειγμα της Βρετανίας όπου από τότε που ε, είχε καθιερώσει το Research Assessment Exercise για τα πανεπιστήμια όταν εφάρμοσε την πολιτική του Λόρδου Σέινσμπορη και του Σερ David King, είδαν εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο στο επιστημονικό output όσο και στον στην οικονομία κλίμακος σχετικά με τα χρήματα που ξοδεύουν. Αυτή τη στιγμή να σας θυμίσω ότι από τα 12 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, τα 6 είναι βρετανικά, ενώ στα 200 καλύτερα 32 είναι ευρωπαϊκά, εκ των οποίων 16 είναι βρετανικά. Άρα πετυχημένα παραδείγματα πολιτικής έρευνας υπάρχουν παντού. Ε, Φυσικά η έκθεση κάνει μερικές σημαντικές και χρήσιμες παρατηρήσεις και συστάσεις για επιμέρους σημεία και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να ενισχύσουμε τον, την αέρα. Φοβάμαι όμως ότι μακροπρόθεσμα αυτά θα αποδειχνούν ανεπαρκή. Εάν εξετάσει κανείς ε, τα δύο κείμενα vis-à-vis, δηλαδή το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται στην ε, σε ζητήματα διοίκησης και στο ίδιο έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον τίτλο «A more research intensive and integrated European Research Area» ε, report που δημοσιεύτηκε το 2008-2009 θα δείτε ότι σε όλα τα κέρια ζητήματα που αναφέρονται στην στρατηγική της Λισαβόνας οι απαντήσεις ως προς την πρόοδο είναι με έναν πολύ ήπιο διατυπωμένο τρόπο, αλλά απλώς είναι αρνητικές. Για παράδειγμα, στην ερώτηση ε, ποια είναι η κατάσταση των πανεπιστημίων στην Ευρώπη σε σχέση με το ε, ερευνητικό τους αποτέλεσμα. Η απάντηση είναι δημοσιεύουν περισσότερο, δεν δημοσιεύουν περισσότερο σοβαρές εργασίες. Έχουμε αυξήσει τις διεθνείς πατέντες. Η απάντηση είναι δεν έχουμε αυξήσει τις διεθνείς πατέντες. Έχουμε ένα consistent σύστημα αξιολόγηση πανεπιστημίων. Η απάντηση είναι δεν έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγηση πανεπιστημίων. Υπό την έννοια αυτή, κύριε Πρόεδρε, θα ήμουν ιδιαίτερο ευγνώμων εάν η στρατηγική της Λισαβόνας και η συνακόλουθη ε, πολιτική που θα ακολουθήσουν μέχρι το 2020 γινόταν αντικείμενο συγκεκριμένης μελέτης σε σχέση με τον λοιπό εξωτερικό κόσμο. Εάν το 2025 η Ευρώπη πρόκειται να αντιμετωπίσει μαζί με την Αμερική την ανατολική θύελα των κρατών BRIC σε σχέση με την έρευνα και την τεχνολογία, θα, ήξερα να ξέρω, να, θα ήθελα να ξέρω πολύ καλά ποια θα είναι η πολιτική μας. Είναι κρίμα επίσης ότι δεν διαβάσαμε σήμερα την έκθεση Μαριμόν και Καρβάγιο, η οποία για πρώτη φορά θέτει τα κύρια ζητήματα. Και τα κύρια ζητήματα είναι πολιτική αριστείας ή πολιτική συνοχής. Η Ευρώπη θα κάνει τα ζητήματά της πιο συγκεντρωμένα, ναι ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Είδα το σφυρί σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβάλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συγγραφείς αυτής της μελέτης. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τις συστάσεις έχετε αναλύσει βασικά τα υπάρχοντα εργαλεία, όμως κατά την άποψή μου για να δημιουργήσουμε ένα άνοιγμα, μια, ένα ποιοτικό ευρωπαϊκό χώρο έρευνα, θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τελείως νέα εργαλεία. Η έκθεση την οποία ανέφερε ο συνάδελφός μας έγινε από μένα και τον κύριο Ράινο Μάμο με βάση τις εμπειρίες που είχαμε όταν είμαστε υπεύθυνοι της έρευνας. Εγώ στην Πορτογαλία, εκείνο στην Ισπανία. Είχαμε κάνει την έκθεση αυτή για τον Επίτροπο Κόντσκι για τη βιοτεχνολογία, για την νανοτεχνολογία. Εξερευνήσαμε όλα τα ε, ε, εμπόδια που υπήρχαν και τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, το οποίο αναφέρθηκε βέβαια, και θα πρέπει να έχουμε καταρχάς έναν στόχο αριστείας και μια ισορροπία. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι ξεχωριστά. Θα πρέπει να δούμε ποια εργαλεία μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, π.χ. Ε, υποτροφίες κτλ. Για να έχουμε τα χρήματα αυτά για την αριστεία και για να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό που ενδεχόμενα να υπάρχει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το Συμβούλιο, το ε, Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας. Μπορείτε να προτείνει Η Ευρώπη μπορεί να προτείνει ένα κοινό, μια κοινή χρηματοδότηση κομισιών κρατών μελών και να γίνει η, αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. national and regional budget to the... Και θα μπορούσε να γίνει μια επιστροφή των κονδυλίων του προπολογισμού σε περιφερειακό επίπεδο για να είμαστε σίγουροι ότι οι περιφερειφέρειες ε, χρηματοδοτούν ε, και κάποιες περιφέρειες οι οποίες δεν είναι τόσο αναπτυγμένες. Και επίσης θα πρέπει να τα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή όταν κάποιος είναι ε, ένας πρώτος ή δεύτερος στην ταξινόμηση, δεν είσαι πρώτος δεύτερος στην περιοχή σου, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι ένα καλό εργαλείο για να ξεκινήσουμε και είναι λιγότερο γραφειοκρατικό όταν συγκρίνεις με το άρθρο 169 γιατί έχουμε τους ίδιους στόχους. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος να απλουστεύσουμε το 169. Αυτά μπορούν να γίνουν παράλληλα, αλλά αυτές οι πανευρωπαϊκές υπηρεσίες πιστεύω ότι διευκολύνουν και η αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αποφύγουμε τον κατακρισμό στην Ευρώπη. Συνάδελφος Τίκαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Λεόν για την παρουσίαση που μας έκανε. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε συνοδεύονται από μια έντονη γραφειοκρατία και πάρα πολλές εταιρείες ε, δεν θέλησαν να πάρουν μέρος σε τέτοιου είδους ε, διαδικασίες. Και ήθελα να ξέρω ποια είναι, ποιο είναι το ποσοστό των project τα οποία υλοποιήθηκαν ε, εκ των υστέρων. Βέβαια, τέτοιου είδους ε, διαδικασίες αναφέρονται σε καινούργιες, σε καινοτόμε ιδέες. Όμως πολλές από αυτές τις καινοτόμες ιδέες ποτέ δεν εμφανίζονται στην αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο την εφαρμοσμένη έρευνα. Επειδή πάρα πολλά χρήματα δαπανώνται για ερευνητικά προγράμματα, πιστεύω ότι θα πρέπει να ευνοήσουμε την εφαρμοσμένη έρευνα. Και ένα από τα ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι το εξή. Γιατί ένα, ένα μεγάλο μέρο αυτών των project δεν υλοποιήθηκαν. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό, δεν υπήρχαν τα χρήματα, γιατί δεν μπορούσαν να ε, εφαρμοστούν πρακτικά. οι ιδέες μπορεί να ήταν καλές, αλλά καλό θα είναι να δούμε ποια ήταν τα εμπόδια τα οποία απέτρεψαν την υλοποίηση αυτών των ε, ερευνητικών ε, project. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώς δεν συμμετέχουν πολύ σε αυτού του είδους τις, ε, τις πρωτοβουλίες. Και το λέω αυτό διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν τα απαραίτητα κονδύλια για την συγχρηματοδότηση. Παραδείγματο χάρη, μια μικρή επιχείρηση, μια μεσαία επιχείρηση, θα πρέπει να ζήσει και για να μπορέσει να επιβιώσει στην αγορά θα πρέπει να ε, αφιερώνει τους ε, βέλτιστους ε, πόρους σε ενέργειες που θα αποδώσουν για την επιχείρηση. Άρα δεν μπορεί να έχει στρατηγικές ομάδες που να ασχολούνται με μακροπρόθεσμα σχέδια τα οποία κάποια στιγμή θα καρποφορήσουν. Δεν υπάρχει δηλαδή επαρκής εγγύηση που να προσφέρεται από αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος να επιτρέπει στις τράπεζες να χρηματοδοτούν κάποια τέτοια προγράμματα. Υπάρχει, υπάρχουν 32 project ε, για αριστεία ε, και πιστεύω ότι αυτή η αναζήτηση της αριστείας θα πρέπει να εμφανίζεται όλο και περισσότερο σε ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεόν. Μπορώ να απαντήσω στα ισπανικά ή προτιμάτε στα αγγλικά. Eh, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους ε, βουλευτές που Πρέπει να τις παρατηρήσεις τους. Πρώτα πρώτα αυτό, σας ευχαριστώ και πάλι. Η έκθεση δεν αποσκοπούσε στο να κάνει μια αξιολόγηση του αντίκτυπου όλων των projects που έχουν γίνει στην Ευρώπη, όλων των προγραμμάτων. Ούτε να κάνει την αξιολόγηση του προγράμματος πλαισίου. Απλώς θέλουμε να σας δώσουμε μια εντύπωση από αυτές τις ε, πρωτοβουλίες. Πολλές από αυτές είναι πολύ πρόσφατες, οπότε και γι' αυτό δεν έχει υπάρξει ακόμα αρκετό χρόνο για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Πολλέ από αυτέ τι πρωτοβουλίε ε, δεν έγιναν καν με, με, ανοιχτού διαγωνισμού ε, που ε, να, να έχουν να έχουν, έχουν, έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επομένω, είναι περίπλοκο το να μπορούμε ακόμα να έχουμε μια συνολική εικόνα και αξιολόγηση του αντίκτυπου. Όμω, μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση σε συγκεκριμένα, μεμονωμένα προγράμματα. Και να σα πω Τρία θέματα από αυτά που αυξηθηκαν είναι σημαντικά. Πρώτα-πρώτα για τα πανεπιστήμια. Θεωρώ ότι η διαδικασία εξονισμού των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων είναι επίσης κομμάτι από την ε, οικοδόμηση του, του, του, της ΕΡΑ. Είναι κλειδί για την Ευρώπη αυτό. Εξού και οι φορείς έρευνας θα πρέπει να εμπλακούν και να μπορούμε να έχουμε κι εμείς μία εικόνα του τοπίου των πολιτικών της γνώσης. Κάτι ευρύτερο από την έρευνα βέβαια. Οπότε χρειάζονται κάποιο είδου μέσα, εργαλεία για να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεταρρύθμιση πανευρωπαϊκά. Και να ληφθούν όμως υπόψη οι που ισχύουν για τα εκπαιδευτικά αυτά ανώτατα ιδρύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αναγκαίο. Δεν έχουμε μηχανισμό αξιολόγησης ε, αυτών των φορέων για αξιολόγηση συνολική. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μόνο ε, σετ ε, κριτηρίων γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα και επικύλα. Τώρα, για τη γραφειοκρατία που μαστίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες προσπαθεί η ίδια η Κομισιόν κάτι να κάνει γιατί από πλευρά των ε, συμμετεχόντων είναι λίγα αυτά τα οποία γίνονται τόσο ώστε να υπάρχει στα στο πλαίσιο πρόγραμμα μια απλούστευση. Όμως για τις πρωτοβουλίες που λέμε τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα διότι σε εθνικό επίπεδο η χρηματοδότηση δίνεται μόνο όταν κανείς υποβάλει προτάσεις και προγράμματα στους εθνικούς φορείς για να μπορέσει να πάρει τα παραπάνω χρήματα τα οποία χρειάζεται. Η διαδικασία αλλάζει από τη μία περίπτωση στην άλλη, από τη μία πρωτοβουλία στην άλλη. Δεν υπάρχει ένας κοινός απλουστευμένος μηχανισμός που να διευκολύνει τις κινήσεις Οπότε η ύπαρξη κάποιων οργανισμών που να μπορούν να έχουν ε, χρήματα από κάποιο, από κάποιο κοινό κορβανά και μπορούσε αυτό να λειτουργήσει σε περισσότερες από μια χώρα θα διευκόλυνε πολύ. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ανέφερε ο τελευταίος από τους πολλαπαν όσον αφορά τη χρηματοδότηση βασική και εφηρμοσμένη. Θα πρέπει να μάθουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν σαν τεχνολογικές και κοινέ ε, δυνάμει του άρθρου 171 έχουν χαρακτήρα που είναι εφηρμοσμένος και αυτό αφορά περισσότερα χαρακτηριστικά τους διότι συνδέονται με, συμφέροντα με ενδιαφέρον από πολλούς κλάδους της βιομηχανίας σε πολλά επίπεδα. Οπότε είναι αναγκαίο και είναι και χρήσιμο να συνδυάσουμε πολύ περισσότερο τέτοιες ε, δράσεις και κινήσεις με άλλες και γιατί να μην συνδυάσουμε μια πρωτοβουλία ή ένα πρόγραμμα ε, στα πλαίσια μιας joint ε, initiative, joint initiative με κάποιο πρόγραμμα του, του τύπου people ή του ιδέα. Και έτσι όλες μας οι κινήσεις και πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες θα έχουν ένα παραπάνω στοιχείο. Θα τις εμπλουτίσει ούτως ώστε να μπορούν να αναγίνουν πιο ελκυστικές στους δυνάμεις συμμετέχοντες. Όπως προελέχθη σε πολλές περιπτώσεις, μπορούμε να στηρίξουμε κάποιους όπως τις ΜΜΕ και αυτό στο πρόγραμμα πλαίσιο ελήφθη σημαντικά υπόψη. Να εξασφαλιστεί ένα κομμάτι σημαντικό, ένα ποσοστό για αυτές τις ΜΜΕ. Όμως, στις πρωτοβουλίες δεν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν αυτές οι κοινέ ε, δομές. Άρα να κάτσουμε να το δούμε αυτό για το μέλλον. Ε, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση, για την συζήτηση, για τις απαντήσεις που δώσατε. Κλείνω το θέμα αυτό λοιπόν της σημερινής διάταξης και προχωρώ στο σημείο 11. για την οδηγία για την καθυστέρηση των πληρωμών. Ο εισηγητή είναι ο συνάδελφο Διάντζελη. Θα ήθελα, ε, σήμερα είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψε, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο κύριε Διάντζελη, να μας κάνετε μια εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά είπατε, πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση, το πρόβλημα της καθυστέρησης των πληρωμών στις ε, εμπορικές συναλλαγές είναι ένα πρόβλημα ε, φοβερά επίκαιρο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βαρύνει την ε, ζωή των επιχειρήσεων και κυρίως την ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλάω για τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα σε οικονομικούς φορείς και ανάμεσα στους οικονομικούς φορείς και την ε, δημόσια διοίκηση. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πολλές ε, πληρωμές καθυστερούν σε σχέση με αυτό το οποίο προβλέπει ή το συμβόλαιο, η σύμβαση ή που προβλέπουν οι, διεθνοί, οι, όροι, οι γενικοί όροι ε, ε, των συναλλαγών η συμβαση η που προβλεπουν οι ώρη οι οροι οι γενικοι οροι των συναλλαγων η οδηγια 35 του 2000 που είχε σαν στόχο τον περιορισμό των, της περίοδου πληρωμών ε, δεν εφαρμόζεται. Και ούτως ή άλλως δεν επιλύει και το πρόβλημα θα έλεγα. Ε, εφτά χρόνια μετά την θέση σε ισχύ της, οι περίοδοι πληρωμών διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλους. Και έχουμε μπροστά μας καταστάσεις πολύ διαφορετικές. Ε, θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματο. 155, 155 μέρες στην Ελλάδα, οι μισές στη Γαλλία, λιγότερες στο Ενωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Επομένως όλη αυτή η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την όλη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ε, θέτει σε κίνδυνο επίσης και την ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για να μην μιλήσω για όλο τον βιομηχανικό κλάδο. Η πρόταση της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή που είναι ένα μέρος των, ενός συνόλου μέτρων που έχουν σαν στόχο την ενδυνάμωση και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για την, για, την, για την έναρξη ξανά των επενδύσεων, για την οικονομική ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη και την παγκόσμια κρίση, ε, θα μπορούσε να δημιουργήσει και νέες θέσεις απασχόλησης. Μετά από αυτή την εισαγωγή, θα ήθελα εν συντομία να κάνω μια συνθετική ανάλυση της πρώτης οδηγίας. Θα ήθελα να διευκρινίσω ευθύ εξ αρχή ότι ο στόχος του κειμένου είναι να εισάγει κάποια στοιχεία ε, ε, ε, Μεγαλύτερη αυστηρότητα και πειθαρχίας ε, μετά την οδηγία 35 του 2000. Και υπάρχει μια πειθαρχία όσον αφορά τις, την περίοδο πληρωμών στις συναλλαγές ανάμεσα στους ιδιώτες και ανάμεσα στους ιδιώτες και στη δημόσια διοίκηση. Καθορίζεται μια, περίοδο, μια προθεσμία 30 ημερών και εδώ επανέρχομαι σε ένα πρώτο θέμα αυτές οι 30 μέρες μένα, αλλά με ένα μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων. Και αυτή η μεγάλη γκάμα των εξαιρέσεων μπορεί να καταστήσει ε, κενή περιεχομένου την διάταξη αυτή. Και κατά την άποψή μου ε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της οδηγίας είναι ο περιορισμός των περιοθωρίων εξαιρέσεων στις, ε, στα συμβόλαια. Θα πρέπει δηλαδή να αποφύγουμε αυτή την, την υπερβολική χρησιμοποίηση των εξαιρέσεων, ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα αποδυναμωθεί τελείω η διάταξη. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε θέματα που αφορούν την αποζημίωση, τις διάφορες ε, ρήτρες που υπάρχουν, ε, η δυνατότητα ε, ίσπραξης των ποσών που δεν αμφισβητούνται και ε, επίσης η... κάτι το οποίο προβλέπει και η οδηγία του 2000 σχετικά με την διατήρηση του, ιδιοκτησιακού καθεστώτος μέχρι ότου και την δυνατότητα κατάσχεσης που υπάρχει μέχρι ότου πληρωθούν κάποια αγαθά και κάποια προϊόντα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι προτάσεις που γίνονται, που έχουν γίνει, ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 87 και απευθύνω μια έκκληση σχετικά με κάποιες πτυχές της οδηγίας. Καταρχάς το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητάτε αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι σε πάρα πολλές χώρες ο ιατρικός και ο νοσοκομιακός τομέας είναι ο τομέας ο οποίος εκτίθεται αν θέλετε περισσότερο, ο οποίος πλήγεται περισσότερο από αυτές τις ε, καθυστερήσεις της πληρωμές από πλευράς τουλάχιστον της δημόσιας διοίκησης και αναφέρομαι και στην ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, στην δημόσια διοίκηση και να συμπεριλαμβάνουμε και κάποιες, υπηρεσίες, κάποιες επιχειρήσεις με μεικτό κεφάλαιο που παρέχουν ε, βασικές πληροφορίες ε, για την, στην κοινωνία. Παραδείγματο χάρη, μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση ε, των συναλλαγών ανάμεσα σε ιδιώτες ή ανάμεσα στους ιδιώτες και στη δημόσια διοίκηση. Αναφέρομαι στα θέματα των προθεσμιών, στα περιθώρια των εξαιρέσεων, στο θέμα της αποζημίωσης για, τις, ε, για τα έξοδα για την, που συνεπάγεται προσπάθεια ίσπραξης, όπως επίσης και μια καταποκοπή αποζημίωση για τις καθυστερήσεις. Ο στόχο υπερημερίας τέλος πάντων. Αυτά είναι μια προκατακτική, μια, μια σειρά προκατακτικών παρατηρήσεων. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την εφαρμογή της, ε, των ε, διατάξεων καταρχάς και αυτό το, για αυτό το σημείο όπως και, για και σε άλλα σημεία χρειαζόμαστε την βοήθεια των, συναδέλφων, από την Επιτροπή χρειαζόμαστε την εμπειρία των κρατών μελών γιατί οι καθυστερήσεις της πληρωμής ε, κινδυνεύουν να παραλύσουν διάφορες, διάφορες, πολλούς σημαντικούς τομείς της οικονομίας μας. Τώρα όσον αφορά τις ημερομηνίες ε, επαφίομαι στις ε, στην Προεδρία. Και ολοκληρώνω λέγοντας ότι ε, οποιαδήποτε ένδειξη και οποιαδήποτε παρατήρηση ε, θα θέλετε να κάνετε σήμερα ή και τις επόμενες μέρες και τις επόμενες εβδομάδες ε, μπορείτε να τις κάνετε και στο γραφείο μου έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε, μια, σε ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο να απαντά με συγκεκριμένο τρόπο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Herzlichen Dank. Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο εισηγητή. Η πρόταση αυτή έχει καθυστερήσει ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τέλος πάντων καλλιόργα παραποτέ παρά ποτέ. Υποστηρίζουμε την ε, έκθεση, αλλά στο άρθρο 5 παράγραφος 4 αναφέρω προ... ε, ζητούμε να ε, υπάρχει ένα maximum 60 ημερών μεγαλύτερη προθεσμία δεν δικαιολογείται και έτσι όπως παρουσιάζονται τα πράγματα εδώ παρά είναι χαλαρά ε, θέλουμε λοιπόν Βεβαίω θέλουμε οι πληρωμές να γίνονται πιο γρήγορα και η πρόταση των 60 ημερών να είναι το maximum. Και εδώ όμω, όταν αναφέρεται αυτό σε κάποιο σημείο παρά είναι χαλάρη η διατύπωση νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει δέσμευση με δημοσιοποίηση με δημοσίευση ορισμένων πραγμάτων. Και τώρα να δούμε τον τομέα business to business μεταξύ επιχειρήσεων, δηλαδή όχι μόνο τη σχέση επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών. Η φιλελεύθερη άποψη θα ήταν ότι αυτά ρυθμίζονται από το δίκαιο των συμβάσεων. Όμως όταν μιλούμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα στο ε, δίκαιο των συμβάσεων και θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να μπουν ειδικοί κανόνες για το τομέα business to business. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, λέει ο πρόεδρος, ο, που, που προέρχεστε από την Δανία, αλλά μιλάτε τέλεια γερμανικά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντω το θέμα των καθυστερήσεων των πληρωμών είναι μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλέ μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης κατά την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα αρχίζει κανείς να αναρωτιέται και για την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών δεν μιλώ για την ανταγωνιστικότητα η οποία επηρεάζεται αρνητικά αλλά μιλάω για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, από εκεί και πέρα αποζημιώσεις στο κήπο ημερίας και τα λοιπά ή, δεν ξέρω αν θα ήταν ε, μέτρα τα οποία θα επέλυναν θα έλυναν το πρόβλημα θα ε, ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το άρθρο 1 παράγραφος 2 παραδείγματος χάρη αναφέρεται η δυνατότητα ε, μάλλον καταργείται η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητήσουν ε, τόκους ή κάτω από 5 ευρώ μετά παρακάτω στο άρθρο 5 για τις, κατα... για τις πληρωμές των δημοσίων υπηρεσιών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε εδώ πιο αυστηροί. Το, ε, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι, οι μη δημόσιες αν θέλετε επιχειρήσεις που όμως παρέχουν κοινοφελείς υπηρεσίε και τα λοιπά αυτές οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να λειτουργούν στις χώρες μας και γι' αυτό θα πρέπει εκεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι ε, ε, 30 με εμείς εδώ θα πρέπει να αγωνιστούμε για τις 30 μέρες, 60 μέρες ίσως είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει βέβαια να καθίσουμε να σκεφτούμε τι θα πει δημόσια επιχείρηση, τι θα πει η μη δημόσια, η μη κρατική επιχείρηση κτλ. Αλλά όταν μιλούμε για 5% του λογαριασμού σαν αποζημίωση αυτά τα 5% ε, θα μπορούσαν να εξαρτώνται από το πότε τελικά έγινε η τελική καταβολή, η τελική πληρωμή. Τώρα για το άρθρο 6 είναι πολύ ε, ασαφής η διατύπωση. Και όσον αφορά τώρα το τομέα business to business, πραγματικά εγώ πιστεύω ότι το δίκαιο των συμβάσεων είναι το βασικό εδώ, διότι μιλάμε για συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Και όταν βλέπουμε από αναλύσεις που έχουν γίνει ότι μεγάλες επιχειρήσεις Ε, πιέζουν τις μικρότερες επιχειρήσεις τότε αυτό είναι άλλο πράγμα δεν είναι θέμα καθυστέρηση πληρωμών Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Νομίζω ότι ακριβώς μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης καλύτερο θα ήταν να ε, εξασφαλίσουμε την ρευστότητα των επιχειρήσεων με τις ε, έγκαιρες πληρωμές παρά να κάνουμε οτιδήποτε άλλο και πραγματικά γι' αυτό η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική τώρα από όταν ε, οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, περιμένουν να πληρωθούν από το δημόσιο ε, δεν μπορούμε να δώσουμε μεγάλες μεγάλα χρονικά περιθώρια εκεί θα πρέπει να αγωνιστούμε τις 30 μέρες πραγματικά οι 30 μέρες είναι το μάξιμο που μπορούμε να δεχθούμε και ε, πραγματικά εγώ νομίζω ότι αν επιμείνουμε τότε θα αυξηθεί η ρευστότητα στην αγορά και θα βοηθηθούν ιδιαίτερα πολύ περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ότι με οποιοδήποτε άλλο μέτρο γρήγορα και αποτελεσματικά λοιπόν θα πρέπει να λειτουργήσουν τα μέτρα αυτά και ε, εάν πάψει να υφίσταται εγκαθυστέρηση των πληρωμών νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο δώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα βεβαίως θα ε, μου πουν ορισμένοι ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στις διάφορες χώρες, ναι ωραία, αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε και το παράδειγμα να το δώσω στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εν συντομία, λέει η κυρία Τόγια, να πω ότι συμφωνώ με τον ε, κύριο Ντεάντζελης, διότι στην, έκθεσή του, ε, στην ομοδότησή του ανάφερε τα βασικά στοιχεία τα οποία έπρεπε ε, να χαρακτηρίζουν ε, ένα τέτοιο κείμενο. Δηλαδή πρέπει να μιλάμε για ε, ευθυκρισία, για συγκεκριμένη εξέταση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας, εφαρμογή του δικαίου και γενικότερα αρχές με τις οποίες είμαστε σύμφωνοι όλοι. Για να υπογραμμίσω ότι είναι σημασία αυτή της διάταξης, να σας πω ότι είναι μία από τις ελάχιστες δεσμεύσεις εκτός από το ΦΠΑ που μας απασχόλησε ε, και είναι από τα αποτελέσματα τα οποία και εμείς σαν πολίτες ε, προωθήσαμε στην προηγούμενη θητεία. Δηλαδή είναι ένα από τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αποφασίσαμε και το περιμένουν ε, το περιμένουμε ιδιαίτερη όλα τα κράτη. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αρχή της, ε, ε, της πειθαρχίας και της δικαιοσύνης που ανέφερε ο κύριος Ντεάντζελ.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 πώς αντιμετωπίζουν οι, οι εκλογείς μας ε, ε, θέματα σαν και αυτά. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά η αγορά. και η Επιτροπή μας σε σχέση με τη συγκεκριμένη γνηματοδότηση πρέπει να ασχοληθεί με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν ε, αυτή της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται δηλαδή για κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και η πείρα μας μας δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Η καθυστέρηση των πληρωμών μπορεί να οδηγήσει σε στην χρεοκοπία πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διότι δεν θα πληρώνονται εγκαίρους. Και το γεγονός ότι υπάρχουν ε, λίγοι βουλευτές εδώ παρόντες στην αίθουσα δεν πρέπει να αποτελεί μια ένδειξη ε, για την σοβαρότητα με την οποία η Επιτροπή μας αντιμετωπίζει το θέμα. Κυρία Μπρίκμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν χαίρεται ιδιαίτερα γιατί άκουσε τον εισηγητή αλλά και τα μέλη της ε, Επιτροπής σας να υποστηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή που είναι ιδιαίτερα ε, σημαντική για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είχε εξαγγελθεί α, μέσα στα πλαίσια του Small Business Act και κάποια υπήρχαν και άλλα στοιχεία ε, παραδείγματο χάρη και ε, ε, η προθεσμία των 30 ημερών που είχε προβλεφθεί και στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας. Ακούστηκαν διάφορα ερωτηματικά για, την, για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Όντως μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά και αυτό που είπατε επίσης για την ε, σημασία μια εναρμόνισης ε, και για τις δημόσιες ε, επιχειρήσεις. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό με τη βοήθειά σας. Υπάρχουν ερωτήματα πιο ουσιαστικά, πιο θεμελιώδη που αφορούν την ελευθερία επίτευξη συμβάσεων. Εμείς βέβαια προβλέπουμε μία εναρμόνιση ε, στις διατάξεις που διέπουν ε, τις, ε, τις συναλλαγές ανάμεσα στο δημόσιο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, διότι εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις και οι συνέπειες είναι πλέον σοβαρές και υπάρχει μια ανισορροπία, δηλαδή δεν υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στους δύο συμβαλωμένους, το δημόσιο από τη μια και τις ιδιωτικές επιχείρησεις από την άλλη. Γι' αυτό είπαμε ότι εδώ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η, η, η, η ελευθερία ε, στην, ε, στις συνδιαλλαγές ε, και αποφασίσαμε να σεβαστούμε και να εφαρμόσουμε την αρχή αυτή στην, στις συναλλαγές ανάμεσα στους ιδιώτες, όχι όμως αδιακρίτως, διότι ε, θέλουμε να, ε, να προστατεύσουμε και τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση κατάχρησης αυτής της ελευθερίας. Προσπαθούμε τώρα να επιλύσουμε τα προβλήματα των της καθυστέρησης των πληρωμών. Ξέρουμε όμως ότι η οδηγία αυτή δεν μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα, διότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για να ρυθμιστεί το πρόβλημα αυτό. Πράγματα τα οποία ε, ξεπερνούν το νομοθετικό πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Θα μπορούσαμε να το, να το εξετάσουμε μαζί σας, να δούμε, ας πούμε, μήπως θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε και να διοργανώσουμε κάποιες εκστρατείες ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος πάντων θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και άλλα μέτρα όχι νομοθετικού περιεχομένου, ε, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τέλος πάντων, είμαστε στη διάθεσή σας και στη διάθεση του εισηγητή να τα, να τα σκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα και να βρούμε τις απαντήσεις που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση εδώ ο συνάδελφος Angelis είπε ότι τον Ιανουάριο θα έχει τέλος του Γενάρη θα έχει έτοιμη τη χνομοδότηση το σχέδιο γνωμοδότης και βεβαίω από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε υποδείξεις και προτάσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε πέντε ακόμη λεπτά στη διάθεσή μας. Σήμερα το πρωί είπαμε θα συζητήσουμε μετά το σημείο 11 της ημερής διάταξης, το σημείο 17, η εισηγήτρια κυρία Τικάου έχει το λόγο για 3,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τον Σκιώδη εισηγητή. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και στους, τρεις, και στους τέσσερις τριλόγους ε, που είχαμε για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Θα ήθελα να κάνω αυτή την παρουσίαση για να Ε, έχω και την δική σας υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με το Συμβούλιο. Καταλήξαμε σε μια αρκετά καλή συμφωνία. Καταφέραμε να διατηρήσουμε τις διατάξεις όσον αφορά τα οικονομικά εργαλεία όχι έτσι όπως τα είχε, τα είχε προτείνει το Κοινοβούλιο, αλλά παρόλα αυτά η Κομισιό μέχρι το 2011 θα αναλύσει τους υπάρχοντες πόρους και θα υποβάλει νέες προτάσεις ε, ή δυνατόν. Σε όλα τα νέα κτίρια από το 2020 θα πρέπει... όλα τα νέα τα νέα κτίρια θα πρέπει να έχουν ε, μηδενικό ενεργειακό, ενεργειακές δαπάνες. Θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε την ενεργειακή απόδοση η οδηγία θα εφαρμοστεί τον, το 2017 και τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν εθνικά προγράμματα και εθνικούς στόχους έτσι ώστε να μετατρέψουν και τα υπάρχοντα κτίρια ε, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία κατανάλωση ενέργειας από το κτίριο αν θέλετε. Τώρα για την κατάρτιση των εμπειρογνωμόνων και για τα πιστοποιητικά της ενεργειακής απόδοσης προβλέπουμε την χρησιμοποίηση της των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακόμα περισσότερο και προβλέπουμε λιγότερες, λιγότερες διοικητικές επιβαρύνσεις έναν ρόλο πιο ε, ενισχυμένο για την Κομισιόν. Η χρησιμοποίηση ε, εφιών ε, ρολογιών, ηλεκτρικών ρολογιών, μετρητών. Υπάρχει και ένα καινούριο παράρτημα επίσης και έχουμε και συγκεκριμένες σαφείς ε, διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε το βέλτιστο κόστος ε, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Αν ένα κράτος μέλος έχει έναν αριθμό ο οποίος να ξεπερνάει κατά παραπάνω από 15% τους ε, αριθμούς, ε, τα ποσά τα οποία έχουμε, τα ποσά αναφοράς, θα πρέπει να υιοθετήσει κάποια διορθωτικά μέτρα. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα καλό κείμενο, το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουμε, πιστεύω. Τώρα θα πρέπει, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με την επιτροπολογία που πρέπει να συζητήσουμε, διότι αυτοί οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται Ε, στις, αρμοδιο... στις συνεργασίες και στις σχέσεις ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνοντας υπόψη για τη συνθήκη της Λισαβόνα. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Χόλ, πολύ πολύ γρήγορα όμως. Θα είμαι σύντομη απλώς να ευχαριστήσω την κυρία Τικάου θερμά, θερμότατα για όλη αυτή τη διαβούλευση και συνεργασία με την οποία ε, χαρακτηρίζεται η συνεργασία της με, με, με, τους ε, σχεδόν ε, αποφασιστικά συνέχισε για τις χειρότερες στιγμές της διαπραγματεύσης όταν νομίζαμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να βγει η συμφωνία τώρα με την Σουηδική Προεδρία και συνέχισε όμως η συγγήτρια να δουλεύει, να προσπαθεί και τα καταφέραμε. Τη αξίζει επομένως ένα μεγάλο μπράβο και αναγνώριση για αυτό που έκανε και επίσης τη αξίζει πλήρης υποστήριξη από πλευράς Επιτροπής των όσων ε, συνέταξε. Τόμος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω τίσω τιμές στην ε, Αντριάννα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό και στον κύριο Φιώνα στον κύριο Κιοντάκη και στο προσωπικό που βοήθησε νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα δεδομένων των δύσκολων διαπραγματεύσεων που ε, έγιναν γιατί πολλές φορές το Συμβούλιο περιχαρακωνόταν γύρω από θέσεις από τις οποίες δεν φαινόταν να μπορεί να μετακινηθεί ε, πιστεύουμε ότι η θα φτάσουμε με, την, με αυτές τις αποφάσεις σε νέα κτίρια τα οποία θα είναι καλύτερα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και τους αρχιτέκτονες, τους πολιτικούς και την κατασκευαστική ε, βιομηχανία και το, τους εμπόρους ακινήτων αν θέλετε ε, όταν είχαμε μια αντίστοιχη ε, νομοθετική πράξη για τις αναπαλαιώσεις ελπίζαμε πολλά εκεί αποτύχαμε αλλά ε, και εκεί το, η, το ακονδύλια που είχαμε δώσει για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας των κτηρίων ήταν μηδενικά. Γι' αυτό και απέτυχε, πέτυχαν τα μέτρα εκεί. Εδώ τώρα λοιπόν ε, ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ε, έχουμε μια ε, ε, έναν αγώνα, μια μάχη να δώσουμε το Μάρτι και έναν αργότερα για επιπλέον κονδύλια που θα πρέπει να πάνε στα κτίρια τα αποτελεσματικά από ενεργειακής απόψεως θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και ιδιαίτερα τον Μάρτιν γιατί πραγματικά αν υπάρχει ένας υπάλληλο της Κομισιόν που δουλεύει με το 40% της ενέργειας είναι ο Μάρτιν. Λοιπόν, δεν είναι... Ε, λογικό να μην υπάρχουν άνθρωποι που θα να δουλεύουν για το θέμα αυτό της ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ ε, για τη συζήτηση όλα τα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε. Κλείνω το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης και πάμε κατευθείαν στην συνεδρία των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Ήδη έχουμε αργήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσει η συνεδρία συντονιστών σε 1,5 λεπτό. Very good. Every, everything on